Υπάρχει αντίσταση λοιπόν που προβάλλεται από τις χώρες που προανέφερα. Γι' αυτό η ρωσική πολιτική αντιμετωπίζει δυσκολίες. Και θα έλεγα ότι γίνεται μια ε, επικίνδυνη αποστολή που δεν μπορεί να πετύχει. Διότι τα ωφέλη του να θεωρηθεί η Ρωσία σαν φυσικό κέντρο, κέντρο μόλου αναπτύξεως του μετασοβιετικού χώρου, αυτά τα ωφέλη όλο και περισσότερο αμφισβητούνται στο μετασοβιετικό χώρο. Όχι σε πασίγνωστες χώρες μόνο όπως η Ουκρανία, αλλά και σε χώρες όπου οι εξελίξεις αυτές είναι νεότερες, όπως η Λευκορωσία. Η όλη διαδικασία της πολιτικής ανάπτυξης του μετασοβιωτικού χώρου είναι περιπλοκότατο θέμα. Και θα έλεγα ότι οι πόροι της Ρωσίας Συνεχίζοντας πάνω σε αυτά που έλεγε ο κ. Λουκιάνοφ, είναι πολύ χαμηλότερη από τις φιλοδοξίες της χώρας αυτής. Και γι' αυτό η επιτυχία μιας τέτοιας πολιτικής είναι πολύ νωρίς να προβλεφτεί τώρα και εγώ δεν θα μπορούσα καθόλου να προβλέψω αν θα πετύχει αυτή η πολιτική ή όχι. Όλων αυτών λεχθέντων εξακολουθώ να συμφωνώ ότι στρατηγικός η Ρωσία και η Ευρώπη χρειάζονται η μία την άλλη, έχουν αντικειμενικό συμφέρον να δημιουργήσουν μια εταιρική σχέση. Και αυτή είναι πολύ δύσκολη αποστολή. Και τώρα, αυτή τη δεδομένη στιγμή, ελάχιστοι αντικειμενικοί αναλυτές θα μπορούσαν να προβλέψουν ταχεία βελτίωση των σχέσεων αυτών. Υπάρχει καμιά φορά ρητή, ε, εκπεφρασμένη επιθυμία από κάποιες χώρες για κάτι τέτοιο, όμως θα έλεγα ότι θα ήταν ακόμα και ανεύθυνο να προβλέψει κανείς ταχείες θετικές εξελίξεις αυτή τη σχέση, διότι υπάρχει μακροσκελής κατάλογος υφισταμένων προβλημάτων σχέση αυτή. Και δοθέντως επίσης ότι οι προσδοκίες, οι πολύ θετικές προσδοκίες που δημιουργήθηκαν αρχές του 2008 και που δημιούργησαν την ατμόσφαιρα για την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη νέα συμφωνία πλαίσιο, όλες αυτές οι προσδοκίες δυστυχώς αλλά και λογικός πως δεν επαληθεύτηκαν με τις εξελίξεις που ακολούθησαν το 2008. Για να αναπτυχθούν με θετικό τρόπο οι σχέσεις αυτές, θα έλεγα ότι δύο πράγματα θα πρέπει να συμβούν όσον αφορά την οτροπία εξωτερικής πολιτικής και της Ευρώπης και της Ρωσίας. Θα πρέπει λοιπόν η Ρωσία να ξεπεράσει την οπορτουνιστική νοοτροπία, να αρπάζει τις ευκαιρίες όταν εμφανίζονται. Αυτή η νοοτροπία αναπτύχθηκε από την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και επειδή η Ρωσία άρχισε να βλέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν έναν φορέα αδύναμο όσον αφορά την εξωτερική πολιτική. Όσον αφορά την Ευρώπη θα έλεγα ότι πριν υλοποιηθεί μια βελτίωση, η Ευρώπη θα πρέπει να αποκαταστήσει την αυτοεκτίμησή της, την αυτοπεποίθησή της στις συναλλαγές της με τη Ρωσία. Αυτή η διαδικασία θα έλεγα ότι λαμβάνει η χώρα, δρομολογήθηκε, πρέπει να αποκατασταθεί λοιπόν η εμπιστοσύνη της Ευρώπης, να ξέρει τι είναι εφικτό σχέση με τη Ρωσία, θα πρέπει να είναι επίμονη η Ευρώπη, θα πρέπει να συνεχίσει πολιτική που βασίζεται ε, στις αξίες και όχι στις ε, σε αφολημιστική βάση, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε αξίες και εκεί διαφοροποιείται η θέση της Ευρώπης από άλλες συμμαχίες στον κόσμο και θα πρέπει να υπομονετική η Ευρώπη και να μην περιμένει μια πολύ ταχεία εξέλιξη. Αυτά και ευχαριστώ για την προσοχή σας. Uh, Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε για την νυφάλια αυτή ανάπτυξη του θέματος. Και οι δύο εμειρογνώμονές μας ξεκίνησαν από το Πανεπιστήμιο της Μόσχας. Μίλησαν βέβαια υπό την ιδιότητά τους ως ειδικών εξωτερικής πολιτικής. Τώρα θα δώσω το λόγο στους πολιτικούς να σχολιάσουν από τη σκοπιά κάποιου ο οποίος δεν αρκείται σε μια περιγραφή ή σε παροχή συμβουλών για μια κατάσταση, αλλά ε, καλείται να λάβει αποφάσεις. Ο κ. Κωνσταντίν Κοζατσόφ. Κύριε Κοζατσόφ, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως πολιτικός ελπίζω να μην σας χαλάσω την συζήτηση, διότι ε, απίλαυσα τις προηγούμενες ε, τοποθετήσεις και ως Ρώσος πολιτικός προσυπογράφω περισσότερα, τα περισσότερα από τα επιχείρηματα που ακούστηκαν τώρα από τους δύο ε, κύριους ομιλητές σας και νομίζω ότι η ανάλυση τους είναι βαθύτερη από μια απλή επιπόλαιη περιγραφή της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής που βλέπουμε καμιά φορά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και σε ορισμένε συζητήσεις όπως η σημερινή. Νομίζω η συζήτηση για τη Ρωσία και την ρωσική εξωτερική πολιτική και τις μελλοντικέ μας σχέσεις πρέπει να γίνεται κυρίως εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με συνομιλητή την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον απλό λόγο ότι εάν αναλύσουμε τις ε, τρεις πρόσφατες κρίσεις του Καυκάσου, την οικονομική και του αερίου, θα δούμε και στις τρεις περιπτώσεις ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδείχθηκε ο πιο ε, αποδοτικός, ο πιο αποτελεσματικός μηχανισμός για την πρόθεση του διαλόγου και περισσότερο από άλλους διεθνείς οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη, όπως το Συμβουλίο της Ευρώπης, όπως το ΝΑΤΟ ή άλλοι. Το καλό νέο είναι λοιπόν ότι υπάρχουν ανοιχτοί, ανοιχτοί διάβλοι διαλόγου σε διάφορα επίπεδα. Πρόσφατα τώρα, χθες, συναντήθηκε η Τρόικα στην Μόσχα. Σήμερα η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα, ενώ το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που επισκέπτεται την Μόσχα μετά από τους σοσιαλιστές που είχαν έρθει τον Νοέμβριο. Αύριο ε, θα αρχίσει ο τρίτος γύρος διαβουλεύσεων για ε, τη νέα εταιρική συμφωνία. Είναι καλό λοιπόν που μένουν ανοιχτοί αυτοί οι διάβλοι διαλόγου και που οδηγούν στο να κατανοούμε ότι μετά την κρίση του Αυγούστου πέρσι, του 2008, δεν μπορεί να συνεχιστεί ε, business as usual, όπως είχαμε πει κατ' επανάληψη στο παρελθόν. Δεν θα πρέπει λοιπόν να είναι τα ίδια τα πράγματα όπως ε, συνήθως, θα πρέπει να γίνουν καλύτερα γιατί χρειαζόμαστε μεν τους στρατηγικούς εταίρους. Το πρόβλημα είναι ότι ούτε η Ρωσία ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν λάβει αποφάσεις σχετικά με το εάν θέλουν να είναι στρατηγικοί εταίροι ή αν θέλουν απλώς να είναι εταίροι, διότι υπάρχει ε, σαφής διάκριση μεταξύ των δύο αυτών όρων. Για μένα, το να είναι κάποιος στρατηγικός εταίρος σημαίνει να μπορεί να λαμβάνει υπόψη και τα συμφέροντα της άλλης πλευράς. Ακόμα και αν διαφωνεί με αυτά. Και ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσουμε να αναπτύξουμε αυτή την στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ ε, Ρωσίας και Ευρώπης που δεν έχουμε ακόμη. Περιγράφοντας τη Ρωσία και την ρωσική εξωτερική πολιτική επιθυμώ να υπενθυμίσω το γνωστό αφορισμό του Winston Churchill ότι η Ρωσία ότι η Ρωσία ποτέ δεν ήταν τόσο αδύνατη όσο θα θέλαμε εμείς στη Δύση και ποτέ δεν ήταν τόσο δυνατή όσο θα ήθελε η ίδια. Παραφράζοντας λίγο αυτό τον αφορισμό θα πω ότι υπάρχουν δύο κατά βάση εσφαλμένες αντιλήψεις οι οποίες εξακολουθούν να επιμένουν εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε χώρες δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός ότι η Ρωσία δεν είναι παρά μία παραλλαγή της Σοβιετικής Ένωσης, ότι εξακολουθεί και είναι εμπειρελιστική, επιθετική και ότι χρειάζεται να βρεθεί κάποιος να τη σταματήσει, να περιορίσει τις δραστηριότητες εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας αν θέλει να αποφύγει τις δυσκολίες. Και η δεύτερη εσφαλμένη αντίληψη, κατά την άποψή μου, είναι ότι η Ρωσία εξακολουθεί να είναι πολύ αδύναμη, δεν διαθέτει επιρροή, ότι κάπου βρίσκεται στη Σιβηρία και καλά είναι να μείνει εκεί. Αυτά μπορεί να ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 90 όταν η Ρωσία πράγματι ήταν αδύναμη και δεν είχε δυνατότητες επιρροής. Γιατί αν ισχύει αυτή η αντίληψη τότε το καλύτερο είναι να αγνοηθεί η Ρωσία μπορεί να έχει κάποια δικά της συμφέροντα, αλλά ας μην μας απασχολεί. Πιστεύω ότι και στις δύο περιπτώσεις οι ερμηνείες αυτές είναι εσφαλμένες. Είναι εσφαλμένη η εικόνα αυτή της σημερινής Ρωσίας. Στη χώρα μου υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ίσως πιστεύουν τα ίδια λιγότερο αφελείς όπως ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 90. Όμως υπάρχουν πολλοί που θα ήθελαν να ξαναδούν τη Ρωσία να εμφανίζεται ως η Σοβιετική Ένωση του σήμερα, ισχυρή στις διεθνείς σχέσεις. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι έχουν πολύ περιορισμένη πολιτική επιρροή στη Ρωσία. Εάν ωστόσο ενισχυθούν η εξήγηση θα είναι ότι η ενίσχυση αυτή που λαμβάνουν προέρχεται μέσα από τις συγκρούσεις οι οποίες προκύπτουν ορισμένες φορές σε σχέσεις με τη Ρωσία και με ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Τέτοιου είδου συγκρούσεις τις χρειάζονται οι ιέρακες και στη Ρωσία αλλά και σε άλλες χώρες οι οποίες έχουν τη διάθεση να αποδείξουν ότι η Ρωσία αποτελεί απειλή για, τα, για τις ευρωπαϊκές κοινέ αξίες και συμφέροντα. Πιστεύω ότι η Ρωσία καλείται να κάνει ορισμένες επιλογές. Είτε θα είναι 100% καθαρή ευρωπαϊκή χώρα, είτε θα είναι κάτι ιδιαίτερο. Γιατί και οι δύο αυτές δυνατότητες υπάρχουν, δηλαδή και συζητούνται και μέσα στη Ρωσία και Νομίζω ταυτόχρονα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται και αυτή να κάνει την ίδια επιλογή. Να αποφασίσει δηλαδή εάν η Ρωσία εντάσσεται στην οικογένεια, στη λέση και είναι καλοδεχούμενη ή είναι κάτι ξεχωριστό. Πιστεύω ότι ένα καλό πρότυπο για τις σχέσεις που μάλιστα έχει αποδείξει την αξία του υπάρχει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Διότι υπάρχουν βασικές διαφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών και σημαντικές. Για παράδειγμα, η θανατική ποινή, τα βασανιστήρια, το Γουαντάναμο, το οποίο βέβαια ε, βρίσκεται καθοδόν για να ρυθμιστεί τώρα, το πρωτόκολλο του Κιώτο και άλλα πράγματα. Υπάρχουν λοιπόν σαφείς ε, διαφωνίες μεταξύ Ευρωπαίων και Αμερικανών, χωρίς όμως να οδηγούν ποτέ σε κανένα τεράστιο πρόβλημα, σε κανένα δηλαδή ανυπέρβλητο εμπόδιο. Αν και στην περίπτωση της Ρωσίας, η αδίποτε διαφωνία αμέσως λαμβάνει διαστάσεις μεγάλου προβλήματος και όπου δεν ε, υφίσταται καμία ανοχή. Γι' αυτό και είναι τόσο σημαντικό τώρα να εξετάσουμε καλύτερα τις μελλοντικέ μας προοπτικές. Γνωρίζω ότι θα έχουμε και άλλη συζήτηση για τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας, αλλά η δική μου ευκαιρία είναι τώρα να μιλήσω και γι' αυτό θα κάνω ένα σύντομο σχόλιο για το σχέδιο εκθέσεως του κ. Ονισκέβιτς, που νομίζω ότι αποτελεί θετική βάση για την περαιτέρω συζήτηση, αλλά είναι απλώς αφετηρία, κατά τη γνώμη μου, γιατί η έκθεση αυτή αναφέρεται κυρίως ε, σε ορισμένε υποδείξεις προς την διαπραγματευτική ομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να πούν υποτιστορισμένα πράγματα στη Ρωσία και για να διορθώσει ορισμένες συμφωνίες με την ε, ε, Ρωσία. Αυτή η προσέγγιση είναι απαραίτητη πράγματι, αλλά δεν είναι επαρκής. Και πιστεύω ότι η έκθεση η οποία θα εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα πρέπει να πάει πολύ περισσότερο σε βάθος και να θίξει τα θέματα, τα προβλήματα της μελλοντική μας σχέσης. Είτε αυτή θα είναι στρατηγική ή όχι. Έχω ακούσει κάποιες φήμες ότι η διαπραγματευτική ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν πρόκειται να δεχθεί τον ορισμό ή ε, τον χαρακτηρισμό στρατηγικού χαρακτήρα δηλαδή για ε, την συμφωνία αυτή, για την ε, συμφωνία αυτή, για την σύμβαση μάλλον αυτή. νομίζω ότι πρέπει να το εξετάσουμε το θέμα γιατί είναι το πιο σημαντικό για τις σχέσεις μας και μόνο εάν επιτύχουμε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό θα, μπορέσουμε να επιτελέσουμε και πρόοδο στις σχέσεις μας που αξίζουν βεβαίως και οι δύο πλευρές. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ λέει και ο Πρόεδρος. Κύριε κάποια σχόλια μονάχα η, το σχέδιο έκθεσης του κυρίου Κέβιτς που είναι ο εισηγητής μας και φυσικά και αντιπρόεδρος της Επιτροπής μας. Ακριβώς είναι μια σύσταση προς το Συμβούλιο. Σύμφωνα με τους κανόνες δεν μπορεί να είναι τίποτα περισσότερο από μια σύσταση. Έχετε σωστή ανάγνωση λοιπόν. Δεν είναι μια γενική έκθεση για τις σχέσεις Ευρώπης και Ευρωπαϊκής Ένωση Ρωσία, Είναι μια συγκεκριμένη σύσταση. Πρωτού περάσουμε τώρα στη συζήτηση. Βλέπετε ότι προσπαθούμε να ακούσουμε τις διάφορες απόψεις των εμπειρογνώμονων, εμπειρογνωμόνων συγγνώμη, και των πολιτικών από τη Ρωσία για να έχουμε μια πιο εμπεριστατωμένη προσέγγιση στην έκθεσή μας. Αλλά είναι γεγονός ότι μετά από τα δύο αυτά κέρια γεγονότα, τον πόλεμο με τη Γεωργία και την κρίση του φυσικού αερίου, έχουμε πραγματικά μια τροποποίηση του πλαισίου, μια μετατόπιση παραδείγματος σε ό,τι αφορά τη σχέση της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θίξατε το ζήτημα της στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Υπάρχουν αμφιβολίες για το κατά πόσον αυτή η σχέση θα πρέπει να λέγεται στρατηγική εταιρική σχέση. Βλέποντας τα πρόσφατα έγγραφα, ψηφίσματα και κείμενα του Κοινοβουλίου, δεν μιλάμε πια για στρατηγική εταιρική σχέση. Ίσως μπορεί να έχει κάποιες σημαντικές πτυχές αυτή η σχέση. Η Ρωσία είναι μια μεγάλη έκταση, αποτελεί το 2% του παγκόσμιου ΑΕΠ, 32% είναι η ευρωπαϊκή οικονομία. Είμαστε 32 φορές μεγαλύτεροι από την Ρωσία. Σε επίπεδο εδαφικό λοιπόν είναι μεγάλη η Ρωσία, σε στρατιωτικό επίπεδο είναι μια μεγάλη δύναμη έχετε 8.000 πυρηνικούς πυράβλους. Λιγότερους έχουμε, δεν έχουμε τόσους πολλούς σίγουρα, δεν ξέρω πόσους, έχουμε. Και χίλιους να είχαμε καλά θα ήταν. Και η τρίτη πτυχή μιας εταιρικής στρατηγικής σχέσης, που για μένα θα είχε μεγάλη σημασία, και βρίσκεται πίσω από τον προβληματισμό σε σχέση με τη Ρωσία ε, σε αυτή τη θητεία του Κοινοβουλίου. Είναι αξιόπιστος εταίρος η Ρωσία, μπορούμε να βασιστούμε σε εσά. Και η κίνηση προς την αλλαγή του παραδείγματος οφείλεται στο ότι η Ρωσία παρεύει τους κανόνες του διεθνούς παιχνιδιού στον πόλεμο με την Γεωργία και επίσης κατά τη διάρκεια της κρίσης για το φυσικό αέριο όπως τονίστηκε από τον Μπαρόζο και τους ανώτατους αξιωματούχους Ευρωπαϊκής Ένωσης που είπαν ότι έγιναν πράγματα τα οποία ήταν απαράδεκτα, η αλλαγή των συνόρων με τη βία και ο μη σεβασμός διεθνώς δεσμευτικών συμφωνιών. Επομένως χρειάζεται να είσαστε και αξιόπιστος εταίρος για να είσαστε στρατηγικός εταίρος. Προφανώς θα θέλαμε να έχουμε μια στρατηγική σχέση με τη Ρωσία θα θέλαμε να μπορέσει να γίνει μια τέτοια επιλογή και από την πλευρά της Ρωσίας που έχει αυτή την τόσο πλούσια ευρωπαϊκή κουλτούρα. Και πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει έτσι να δει την Ρωσία ως ένα εταίρο και σύμμαχο ο οποίος συμμερίζεται τις ίδιες αξίες με μας. Σίγουρα η ελίτ, η πολιτική και η οικονομική είναι τμήμα των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά πάντως που άκουσα από τους εμπειρογνώμονες εξ ευωνίμων και επίσης από τα σχόλια του Κοσατσόφ είναι περισσότερο για το τι δεν είναι η Ρωσία. Εμείς περιμένουμε να δούμε μια απάντηση για το ερώτημα τι είναι η Ρωσία. Και γι' αυτό θα θέλαμε να έχουμε πιο συγκεκριμένες εικόνες, γιατί υπάρχουν πολλές παρανοήσεις, πολλές λανθασμένες εικόνες και αντιλήψεις για τη Ρωσία. Ας προσπαθήσουμε να έχουμε επακριβείς αντιλήψεις και εικόνες για τη Ρωσία και ελπίζω ότι αυτή η συζήτηση θα μας βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή. Οχτώ ομιλητές έχω τώρα στον κατάλογο. Θέλω να χαιρετήσω την Ρία Όμεν Ρέιτεν, που είναι επικεφαλής της ε, αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την Ρωσία και θα της δώσω και τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ καλό που σήμερα διεξάγεται αυτή η συζήτηση διότι γνωρίζουμε ότι χρειαζόμαστε ένα τον άλλον και χρειαζόμαστε ένα στατικικό εταίρο, δηλαδή τη Ρωσία και η Ρωσία χρειάζεται εμάς σαν στρατηγικό εταίρο. Αυτή είναι η αφετηρία μου. Αυτή που χρησιμοποιώ και σε άλλες επαφές που έχω με τη Ρωσία. Λοιπόν, Πρόεδρε, αν μιλάμε για μια στρατηγική εταιρική σχέση, θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι μαζί ότι υπάρχουν παρεξηγήσεις και από την πλευρά μας και από την πλευρά της Ρωσίας, λανθασμένες εικόνες. Αν δεν το δούμε το θέμα και από τις δύο πλευρές, δεν θα μπορέσει να προχωρήσει αυτή η στρατηγική εταιρική σχέση. Και όπως είπαν οι ομιλητές, έχουμε διαφορετικό παρελθόν όλοι μας και θα πρέπει να συνηθίσουμε το νέο μέλλον που θα έχουμε όλοι μαζί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι ξεκινά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δημιουργεί σχέσεις με τις γύρω χώρες και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, 27 χώρες, έχουμε αυτή την ισχύ. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ισχύ, ούτω ώστε να δημιουργήσουμε καρποφόρες σχέσεις με τους άλλους. Αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική αφετηρία. Για πιο συγκεκριμένα θέματα, ξέρω ότι περνάμε μια τεράστια οικονομική κρίση όλοι. Όχι μόνο εδώ, αλλά και στη Ρωσία. Δεν ξέρω πού είναι μεγαλύτερος ο αντίκτυπος. Θα ήθελα να ξέρω όμως ποιες είναι οι πολιτικές συνέπειες. Τι επεξεργάζεστε τι μπορούμε να κάνουμε από κοινού, πώς μπορούμε να ενισχυθούμε στις προσπάθειες που καταβάλουμε. Πρόεδρε, νομίζω ότι στην έκθεση του κύριου Ονισκίεβιτς είναι πολύ σημαντικό να δούμε ποιοι τομείς πολιτικοί και πρακτικοί τομείς μπορούν να μας βοηθήσουν για να συνεργαστούμε με τη Ρωσία. Χρειαζόμαστε αυτή τη συνεργασία για να ξεπεράσουμε αυτή την οικονομική κρίση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, κυρία μου. Και τώρα ο κ. Ονισκίεβιτς, ο συγγητής, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Καταρχάς, θα ήθελα να πω μερικά λόγια για την έλλειψη ιδεολογίας πίσω, πίσω από τη συμπεριφορά της Ρωσίας και τη θέση της Ρωσίας. Αληθεύει. Όμως υπάρχει και κάποια ιδεολογία που θα μπορούσε αυτή να περιγραφεί ως η προώθηση της μη φιλελεύθερης δημοκρατίας. Δηλαδή δημοκρατίας που περιορίζεται μόνο στους εκλογικούς μηχανισμούς ε, και αρνιέται την ανάγκη να υπάρχει ένα θεσμικό σύστημα ελέγχων και ισορροπιών. Και όλη η συμπεριφορά της Ρωσίας στο διεθνές προσκήνιο, οι στενές σχέσεις με τη Βενεζουέλα και ένα φλερτάρισμα με την Κίνα ίσως δημιουργούν την εντύπωση ότι η Ρωσία δεν ακολουθεί συγκεκριμένη αποστολή να διαδώσει αυτή την προσέγγιση. Αλλά θέλει να ενοποιήσει παρόλα αυτά χώρες που έχουν παρόμοια πολιτικά συστήματα και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Ίσως μπορεί να συζητήσει κανείς σε ποιο βαθμό αυτό έχει σημασία και πώς θα διαμορφώσει αυτή η προσέγγιση στο μέλλον. Δεύτερον, το πρόβλημα της στρατηγικής εταιρικής σχέσεως και η χρησιμοποιούμενη ορολογία. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι η σχέση με κάποιον μπορεί να ονομάζεται εταιρική σχέση από τη στιγμή που μοιραζόμαστε αρκετές κοινέ αξίες. Και εδώ τίθεται το θέμα. Με τη Ρωσία έχουμε προβλήματα στον αφορά τις κοινέ αξίες. Με τη Ρωσία όμως έχουμε στατηγικά συμφέροντα κοινά. Εγώ θα αντέστρεφα το όλο ζήτημα. Έχουμε κάποια στατηγικά κοινά συμφέροντα με τη Ρωσία. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες απαριθμώντας κάποιο κατάλογο. Θα μπορούσε όμως να υποβληθεί συγκεκριμένος κατάλογος τέτοιων συμφερόντων. Τέλος, ε, να επιστρέψω στο δόγμα Πούτιν-Μεντιέντεφ ε, που δημιουργεί κάποιες ε, ανησυχίες. Ποια είναι η ιδέα πίσω από το δόγμα ότι η Ρωσία μπορεί να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των πολιτών της όπου βρίσκονται αυτοί και για την άμυνα αυτή να χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα. Αυτό είναι κάτι που ανησυχεί κάπως. Και είδαμε τι έγινε με τη Γεωργία και κυρίως την Αυχαζία. Και είναι σημαντικά αυτά που συμβαίνουν. Διότι οι δράσεις στην Αυχασία είναι διαφορετική από, ότι, από αυτά που έκανε η Ρωσία στη Νότια Οσετία, διότι στη Νότια Οσετία σε κάποιο βαθμό η Ρωσία μπορούσε να ισχυριστεί ότι αντέδρασε στη στατιωτική επέμβαση της Γεωργίας στη Νότια Οσετία. Η επέμβαση στην Απχαζία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, είναι σαφής περίπτωση προληπτικής στατιωτικής δράσης. Διότι αυτό μπορεί να δημιουργεί την εντύπωση ότι η Ρωσία μπορεί να εισαγάγει στην πολιτική της συμπεριφορά αυτό το στοιχείο. Και αυτό ανησυχεί. Τέλος. Ο κ. Κοσατσόφ σωστά είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή θα πρέπει να καθορίσει τη σχέση της με τη Ρωσία θα ανήκει στην ίδια οικογένεια η Ρωσία ή όχι. Όσον αφορά την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ρωσία δεν θέλει να είναι υποψήφια χώρα από ό,τι καταλαβαίνω και είναι φυσικό βλέποντας αυτά που λέει ο πρόεδρος Πούτιν ότι είτε πρέπει να είναι πλήρως κυρίαρχη και ανεξάρτητη η Ρωσία ή να μην υπάρχει καθόλου. Αν μια χώρα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκχωρεί κάποιο τμήμα της κυριαρχίας σε υπερεθνικούς θεσμούς. Οπότε δεν ταιριάζει με την ιδέα της διατήρησης του 100% της ρωσικής κυριαρχίας. Ευχαριστώ κύριο Σκίεβιτς και τώρα κύριος Ρότσεκ, Αντιπρόεδρος Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. I have more than... Ε, μάλλον ερωτήσεις έχω να κάνω εγώ και όχι σχόλια. Είπαν ότι Δεν υπάρχει κανένα σύστημα ασφάλειας στην Ευρώπη που να το εμπιστεύονται όλοι οι συμμετέχοντες. Πώς βλέπει ε, ο κύριος Λουκιάνοφ το ε, σύστημα που έχουμε τώρα. Θεωρεί ότι δεν είναι το σωστό πλαίσιο. Η ερώτησή μου δηλαδή έχει το νόημα. πώς ε, ε, βλέπετε τη μελλοντική αρχιτεκτονική αυτού του συστήματος, δηλαδή ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος του ΆΣΕ, ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος ε, του ΝΑΤΟ. Για την ώρα υπάρχει το ΝΑΤΟ που βέβαια συμμετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς. Πώς θεωρείτε λοιπόν ότι η μελλοντική αυτή αρχιτεκτονική ενός συστήματος ασφαλείας θα έπρεπε να είναι ώστε να το εμπιστεύονται όλοι, επομένως όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η Ρωσία και βέβαια οι χώρες οι οποίες βρίσκονται ανάμεσα στους δύο αυτούς πόλους ε, Ένωσης και Ρωσίας. Η δεύτερη ερώτησή μου είναι η εξής. Λέτε ότι κάποια, κάποιο είδους συμφωνία συνολική που θα έπρεπε να περιλαμβάνει όλες τις πτυχές των σχέσεών μας φαίνεται αδύνατη για την ώρα. Ρωτώ λοιπόν ποιο δρόμο να επιλέξουμε για να προχωρήσουμε. και μέσα στα πλαίσια της παρούσας οικονομικής κρίσης αλλάζει συνεχώς η κατάσταση και στην ε, Ρωσία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο παγκόσμιο επίπεδο. Αν δεν έχουμε λοιπόν ένα ξεκάθαρο ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο να ρυθμίζει και τις σχέσεις μας θα ε, προκύψουν περισσότερα προβλήματα παρά ε, καλά πράγματα. Αν μπορείτε να πείτε λίγα λόγια και γι' αυτό δηλαδή. Ευχαριστώ. Ο σας ευχαριστώ και εγώ. Ένα σχόλιο, δύο ερωτήσεις. Σχόλιο. Αμέσως μετά την δείξη του ψυχρού πολέμου, η σφαίρα επιρροής της Σοβιετικής Ενώσεως στην Ανατολική Ευρώπη εξαφανίστηκε και μας επέτρεψε σε εμά να μπούμε πλέον ανεξάρτητα και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν τω μεταξύ η Ρωσία έκανε ένα πολύ ισχυρό comeback και κυρίως ε, από το 2000 και μετά άρχισε να αμφισβητεί τις παλές συμφωνίες οι οποίες, ε, τις οποίες είχε διαπραγματευτεί η Ρωσία στη δεκαετία του 1990 και ζητεί νέες συμφωνίες οι οποίες να απηχούν αυτή τη νέα ισχύ της Ρωσίας και τον ρόλο που θεωρεί ότι πρέπει να παίζει ε, στη λήψη αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Το ερώτημα είναι αυτή η επιστροφή της Ρωσίας συνοδεύεται ή όχι από μια προσπάθεια να επανοικοδομήσει τη σφαίρα επιρροής που διέθετε η οχι απο μια προσπαθεια να επανικοδομησει τη Ένωση στην Ανατολική Ευρώπη. Και παρά το γεγονός ότι τώρα πλέον οι χώρες μας είναι μέλη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Εάν πάρετε το γεγονός για παράδειγμα ότι αυτοί που επλήγησαν περισσότερο, αυτές που επλήγησαν περισσότερο οι χώρε που πλήγησαν περισσότερο, για παράδειγμα, από την διακοπή του φυσικού αερίου ήταν ακριβώ εκείνε οι χώρε. Τα νέα μέλη δηλαδή των, νέων, των δύο αυτών διεθνών οργανισμών και έγινε και μια προσπάθεια να ε, συγκληθεί μια διάσκεψη κορυφή για το φυσικό αέριο στη Μόσχα υπό τι ε, συνθήκες αυτές και ε, βέβαια οι χώρε αυτέ θα ήταν υποχρεωμένε να πάνε στη Μόσχα αφού από εκεί προέρχεται το αέριο Υπάρχει έντονο συμβολισμός δηλαδή. Και υπάρχει και η προσπάθεια πλευράς Ρωσίας να πιστούν οι παλές χώρες μέλη να συμπεριφέρονται στις νέες χώρες μέλη σαν μια ειδική κατηγορία ώστε έμεσα να επιτρέψουν στην, στην ε, Ρωσία να συνεχίσει να έχει λόγο ε, στα πολιτικά τους πράγματα. Αυτό το σχόλιο το κάνω ως πλαίσιο για να κατανοήσετε τις ερωτήσεις μου. Πρώτη ερώτηση, πώς διατηρεί την ισορροπία η Ρωσία στη σχέση της με την Δύση, ας πούμε έτσι, μεταξύ άμεσων σχέσεων με ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση ως οργανισμούς και σχέσεις με επιμέρους χώρες μέλη. Ποια από αυτές τις σχέσεις είναι πιο σημαντική ή ποια θα διαμορφωθεί ως πιο σημαντική στο μέλλον. Δεύτερο, υπάρχει μια βιασύνη από πλευράς Ρωσίας να επωφεληθεί όσο το δυνατόν περισσότερο από την πρόσφατη ισχυρή της θέση. Αν όμως αναλύσουμε τις τάσεις σε σχέση με τα αποθέματα αερίου, την υποδομή κτλ. Βλέπουμε στην ουσία ότι φαίνεται να πλησιάζει πλέον στο αποκορύφωμα, διότι εάν δεν συνεχίσουν να υπάρχουν επενδύσεις κτλ. σε αυτούς τους τομείς, από εκεί πέρα θα αρχίσει μια <clears throat> πτώση μια αυθύνουσα πορεία της Ρωσίας. Πώς το βλέπετε αυτό για το μέλλον. Ευχαριστώ κύριε Πάσκο. Ο κύριος Γκάλερ, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα στον κύριο Κόζατσεφ. Η οικονομική κρίση έδειξε ότι και στη Ρωσία τα έσοδα από την πώληση φυσικών πόρων έχουν μειωθεί δραματικά και επομένως με τον τρόπο αυτό δεν έχουν αρκετά χρήματα για να επιδοτήσουν κάποιες ε, βιομηχανίες, κάποιες δραστηριότητες οι οποίες χρειάζονται οπωσδήποτε εξυγχρονισμό και είναι υποχρεωμένοι να συνεχίσουν να λειτουργούν με τις παλιές δομές. Παρά το γεγονός θα ήταν πολύ καλύτερο να είχαν εξυγχρονιστεί αυτές οι δομές. Λόγω αυτού του γεγονότος τώρα. το γεγονός ότι όλοι αυτοί η στρατηγική τομείς δεν είναι τομείς συνεργασίας με τη Δύση πια. έχει λεχθεί ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε ξένους επενδυτές γιατί είναι τομείς στρατηγικής σημασίας. Είναι αυτό κάτι το οποίο είναι παραγωγικό, μήπως θα χρειαζόταν περισσότερη συνεργασία με την ευρωπαϊκή οικονομία για να εξασφαλίσετε αυτό τον εξυγχρονισμό στις ε, βιομηχανία σας και για να εξέλθετε και από την κρίση μεταξύ άλλων. Ευχαριστώ ο κύριος Σβόμποντα, αντιπρόεδρος των Σοσιαλιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω ένα σχόλιο και ένα ερώτημα. Καταρχήν θέλω να αναφέρω δύο προϋποθέσεις που πιστεύω ότι είναι απαραίτητες για να έχουμε μια εταιρική στρατηγική σχέση. Μία που αφορά την ευρωπαϊκή πλευρά, μία τη ρωσική πλευρά. Από την ευρωπαϊκή πλευρά δεν μπορούμε να έχουμε στρατηγική εταιρική σχέση αν σε οποιαδήποτε κρίση λέμε φταίει η Ρωσία. Παράδειγμα είναι η ενεργειακή κρίση. Δεν είναι γεγονός ότι η Ρωσία δεν έδρασε με τρόπο ο οποίος ήταν υπεύθυνο. Το Συμβούλιο και η Κομισιόν μπορούν να πούν ότι <clears throat> και οι δύο πλευρές είναι υπεύθυνε για την κρίση και η Ουκρανία έπαιξε ρόλο και ανέλαβε ευθύνε στην περίπτωση τη κρίση για το φυσικό αέριο. Είναι απαραίτητο να έχουμε μια ισορροπημένη αντιμετώπιση και χαίρομαι για αυτά που είπε ο κ. Σονισκέβη για τι διαφορέ στην αντιμετώπιση τη Νότια Οσετία και τη Απχαζία. Υπάρχουν διαφορέ. Αν δεν δούμε αυτέ τι διαφορέ και έχουμε μια μονολυθική αντιμετώπιση που είναι ότι η Ρωσία φταίει για όλα, αυτό δεν νομίζω ότι αποτελεί βάση για τη δημιουργήση και την οικοδόμηση μιας στρατηγικής εταιρική σχέση, Από την, την άλλη πλευρά όμω, και η Ρωσία θα πρέπει να σκεφτεί καλύτερα τη σχέση της για την κοινή γειτονία τη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και πώ θα αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να επεκτείνει την επιρροή της βεβαίω. Αλλά αυτό θέλουμε να το κάνουμε προσφέροντας κάτι. Κονδύλια, καλή συνεργασία, δυνητικότητα ένταξης. Ενώ από την άλλη πλευρά η Ρωσία δεν έχει βρει κάποιους εποφελείς τρόπους να διατηρήσουν ή να επεκτείνουν την επιρροή τους προσφέροντας κάποια θετικά στοιχεία. Εδώ βρίσκεται το πρόβλημα για μένα και εδώ θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει ένας ειρηνικός ανταγωνισμός, μια ειρηνική άμυλα προσφοράς ωφελημάτων στους γείτονές μας και αυτό ίσως είναι προϋπόθεση για να μπορέσει η Ρωσία να συμμετάσχει σε μια στρατηγική εταιρική σχέση, γιατί αυτό θα οδηγήσει και σε μια μορφή συνεργασίας. Για τον κύριο Μόσες τώρα, <clears throat> είπε ότι οι γειτονικέ της χώρες δεν θέλουν να έχουν ακόμα τη Ρωσία που ήταν το κέντρο της Σοβιετικής σφαίρας. Στην Ουκρανία βέβαια υπάρχουν διχασμένες απόψεις, αλλά τι γίνεται στο Καζακστάν και το Αζερβαϊτζάν, αν μπορείτε να κάνετε μια παρουσίαση για το αν αυτή είναι η ίδια θέση όλων των χωρών ή αν υπάρχει μια διαφοροποίηση μεταξύ των γείτονων της Ρωσίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σβόμποντα, μου αρέσει αυτή η έννοια του ανταγωνισμού γεωνοδορίας. Ας ταξιδέψουμε προς Νότον, Νότιος Κάφκασος, η κυρία Σλέρ Μπεγκέν είναι πρόεδρο τη αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον Νότιο Κάφκασο και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα μιλήσω γαλλιστή αν επιτρέπετε. Ευχαριστώ του ομιλητέ για τι παρεμβάσει τους που μας διαφωτίζουν αλλά που μας αφήνουν και κάπως πεινασμένους για συνέχεια. Θα ήθελα να πω προς τον κύριο Καζουτσέφ ότι όλα δεν είναι τόσο αρνητικά όσον αφορά τις σχέσεις και όταν αναφερθήκατε στο πρωτόκολλο του Κιώτο η έννοια ήταν αντίθετη. Δεν υπέγραψαν οι ΙΠΑ το πρωτόκολλο του Κιώτο και τους κατηγορήσαμε γι' αυτό. Αντίθετα το υπέγραψε η Ρωσία και χάρη στην υπογραφή της Ρωσίας το πρωτόκολλο του Κιώτο ε, μπόρεσε να ε, προωθηθεί. Ήταν θετική συμφωνία. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στην όλη δομή της προσέγγισης. Κάτι οικοδομείται, δεν ξέρουμε αν υπερβολικό ή όχι αυτό που οικοδομείται. Ο κ. Σονεσκίβης είπε κάποια πράγματα αναφερθήκατε σε κοινέ αξίες. Τις έχουμε αυτές τις κοινέ αξίες και θεωρούμε ότι μοιραζόμαστε αυτές τις κοινέ αξίες της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τη Ρωσία. Το ερώτημα που θέτω είναι σήμερα υπάρχει κάποια εξέλιξη όσον αφορά τη δημοκρατία, διότι βλέπουμε πολύ καλά ότι οι διάφορες πλευρές διεκδικούμε τη δημοκρατία, όμως υπάρχει κάποια εκτίμηση της δημοκρατίας αντίληψη δημοκρατίας Άλλη αντίληψη Ρωσία, άλλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, άλλη στι Αφρικανικέ και σαλαβικές χώρε. Υπάρχει ένα νέο ορισμό τη δημοκρατία που διαμορφώνεται. Μπορούμε να διαρωτηθούμε. Και όσον αφορά αυτή τη δημοκρατία, την έννοια δημοκρατία. Πώ επιβάλλεται η δημοκρατία, με τη σύγκρουση. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τις συγκρούσεις αυτές του Αυγούστου μεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας και θέτω το ερώτημα στον κύριο Μωυσέ. Αναφερθήκατε σε χώρες πελάτες, σε ζώνες επιρροής. Σήμερα τι είναι αυτές οι ζώνες επιρροής. Πώς το εξηγείτε εσείς ότι μια χώρα που έχει κοινέ αξίες που τις μοιράζεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης με άλλες χώρες επιτρέπει στον εαυτό της να εισβάλλει σε τέτοιο μεγάλο βάθος στη γειτονική χώρα που είναι πολύ μικρή χώρα σε σχέση με την πολύ μεγάλη ισχύ της ε, Ρωσίας. Προσπαθούμε να καταλάβουμε εμείς τι σημαίνει ζώνη επιρροής. Όταν βλέπει κανείς ότι η Ρωσία πρότεινε στην Νότια Οσετία και στην Απχαζία την εγκατάσταση στρατιωτικών βάσεων και στρατιωτικές βάσεις της Νοτιού Οσετίας θα είναι στα 30 με 40 χιλιόμετρα απόσταση από την Τυφλίδα, Μπορεί να καταλάβει κανείς ότι αυτή η μικρή δημοκρατία δεν αισθάνεται καθόλου ασφαλής πια. Πώς μπορείτε να το εξηγήσετε αυτό για να μπορέσουμε και εμείς να καταλάβουμε τη Ρωσία και τι σημαίνει εν τη αυτή περιπτώσει η ασφάλεια μιας χώρας. Είμαστε στα πλαίσια πολιτικής γειτονίας, δεν είναι πολιτική γειτονίας με τη Ρωσία και με τις χώρες του Καυκάσου και με την Τουρκία. Αλλά σε αυτό το πλαίσιο δεν μπορούμε να ελπίζουμε να έχουμε πολιτική καλής γειτονίας σε ένα άμεσο μέλλον μέσα από τα πλαίσια που προανέφερα. Ευχαριστώ κυρία Ισλερ Και τώρα ο κύριος Λάξ από τους ε, φιλελευθέρους έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρο, κύριε Πρόεδρε συγγνώμη και ευχαριστώ και τα μέλη του πάνελ για τις παρεμβάσεις τους. Τις εξετίμησα άλλος ιδιαίτερος. Έχω δύο ερωτήσεις λίγο πολύ παρόμοιες με τις ερωτήσεις της κυρίας Όμεν Ράιτεν και σχετίζονται και κατά πολύ με αυτά που είπε ο κύριος Γκέλλερ. Στο άμεσο μέλλον, οι συνέπειες της πολύ μεγάλης οικονομικής ύφεσης στη Ρωσία, ποιες θα είναι. Διότι συζητάμε μέσα σε ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο. Αλλά για να ξεκινήσουμε, πρέπει να δούμε τι γίνεται εδώ και τώρα. Οι Ρώσοι ηγέτες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με την ύφεση, από ό,τι καταλαβαίνω. Το ερώτημα είναι τι αντίκτυπο θα έχει αυτό στην πολιτική. Οι ηγέτες θα θέλουν περισσότερο κοινέ λύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή λιγότερες. Θα γίνει ισοστρεφής η Ρωσία γινει εσωστρεφης επιθετικά εξωστρεφής. Αυτό είναι το ερώτημα. Το πρώτο. Το δεύτερο ερώτημα. Με ποιο τρόπο ή υπάρχει τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να συμβάλλει στην επίλυση των οικονομικών προβλημάτων και να βοηθήσει τη Ρωσία να ξεπεράσει την οικονομική κρίση. Κύριος Ντουκαζόλιομι με από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα, λέει και ο Ντούκα Ζόλιομι. Ακούσαμε ενδιαφέρουσε ε, παρουσιάσεις. Νομίζω ότι είναι σημαντική συνεδρίαση, διότι αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα, πρέπει να κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, σχετικά με τις παρουσιάσεις, ένας από τους ομιλητέ είπε ότι η Ρωσική Ομοσπονδία δεν είναι μια νέα μορφή της παλιάς Σοβιετικής Ενώσεως και δεν είναι υπεριαλιστική. Τι είναι μια μεγάλη δύναμη που δημιουργεί τη ζώνη επιρροής της και προστασία συμφερόντων της. Αν δούμε τις πρόσφατες εξελίξεις, είδαμε δύο σημαντικά γεγονότα, τον πόλεμο Ρωσίας-Γεωργίας, τη σύγκρουση στον Κάφκασο και την ε, κρίση του φυσικού αερίου. Προσετέθηκε η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση. Και εκεί η Ρωσία έδειξε τι έχουν υπόψη τους σαν ζώνη επιρροής στη μετασοβιετική εποχή. Πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα όσα συνέβησαν στον Κάφκασο, πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε τη συμφωνία που συνήθιγε η αεροπορική συνεργασία με τον Λουκασένκο τις διάφορες αυτές συμφωνίες που συνήθισαν και την αποχώρηση κάποιων ε, ξένων δυνάμεων, αμερικανικών δυνάμεων. Η κυρία Ισλέρ Μπεγκέν αναφέρθηκε σε έναν τομέα που με ενδιαφέρει. Η σύγκρουση στον Κάφκασο και τα προβλήματα στον Κάφκασο δεν έχουν επιληθεί. Υπήρξε συμφωνία κατά πάψος του πυρός. Αλλά στα σημεία, τα σημεία 5 και 6 της συμφωνίας ε, δεν υλοποιήθηκαν. Το σημείο 5 αναφέρεται στην επαναφορά στην προπολεμική κατάσταση. Άρα πρέπει να επανέλθουμε στην κατάσταση που επικρατούσε μετά τη συμφωνία του 1991 και ο αριθμός των θετικών δυνάμεων των στατιωτών. Έχουμε αρκετές χιλιάδες όμως Ρώσους στατιώτες. Έχουμε εγκατάσταση ε, στρατιωτικών βάσεων ρωσικών Πώς μπορεί να υπάρξει αξιοπιστία. Πώς μπορούμε με κάποιον μη αξιόπιστο εταίρο να δημιουργήσουμε μια στατηγική εταιρική σχέση. Απλή, έστω και απλή εταιρική σχέση. Πολλό μάλλον δε μια στατηγική, εταιρική σχέση. Η κυρία Ισλέρ Μπεγκέν αναφέρθηκε ε, σε κοινά συμφέροντα, κοινέ αξίες. Ε, για μας οι κοινέ αξίες είναι καθαγιασμένες, δηλαδή συμμόρφωση με, τις, με τα ανθρώπινα δικαιώματα, προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στη Ρωσία παραβιάζονται καθημερινά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το δικαίωμα να εκφράζεται κανείς ελεύθερα, η ελευθεροτυπία, όλα αυτά παραβιάζονται. Άρα είναι λέ, δύσκολο να βρούμε κοινέ αξίες ε, για να πετύχουμε μια σοβαρή εταιρική σχέση. Αυτό πιστεύω. Θέλουμε μια σοβαρή σχέση, ούτε στρατηγική ούτε απλή, λέει ο πρόεδρο. Ο κ. Ματσάκη. έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παρόλε τι τρέχουσε διαφορέ μα Παρόλες τις τρέχουσες διαφορές μας με τη Ρωσία, έχουμε και πολλά κοινά στοιχεία. Και οι μεν χρειαζόμαστε τους δε. Παρά το γεγονός ότι τα παλαιότερα σύννεφα στον ορίζοντα. Εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε με τους δε. Κάποια στιγμή πρέπει να συμφωνήσουμε. Και για μένα η φυσική πορεία θα είναι της Ρωσίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια αυτό είναι ένα όραμα για το μέλλον. Διερωτώ με κατά πόσο ο ρωσικός λαός και οι ρώσοι πολιτικοί έχουν και αυτοί ένα τέτοιο όραμα και αν είναι διατεθειμένοι να εργαστούν προς την κατεύθυνση αυτή, ίσως να κάνουν αλλαγές, να κάνουν θυσίες, αλλά να κινηθούν προς την κατεύθυνση μιας ένταξης. Δεύτερο, και μιλώντας για εμπιστοσύνη, χρειάζεται να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη μεταξύ μας. Και το να διαθέτει κανείς 8.000 ε, πυρηνικές κεφαλές ή 7 και 6.000 δεν βοηθεί στο να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη. Διερωτώ λοιπόν, κατά πρώτον, τι τις θέλει όλες αυτές τις πυρηνικές κεφαλές στην Ευρώπη η Ρωσία. Τι φοβάται η Ρωσία. Τι θέλει, τι, τι της χρειάζεται 8.000 πυρηνικές κεφαλές. Υπάρχει άραγε τρόπος η Ρωσία να μπορεί να μειώσει σημαντικά τον αριθμό αυτών των κεφαλών, ώστε να δείξει κιόλας ότι εμπιστεύεται την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εταίρους. Τέλος, αυτή η σχέση για την ειρήνη. Ποιος είναι ο ρόλος της Ρωσίας μέσα σε αυτήν. Έχει σκοπό, έχει φιλοδοξία να παίξει ένα σημαντικό ρόλο μέσα σε αυτήν ή όχι. Η πρόταση για να ενταχθεί η Ρωσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχεται την Κύπρο, ε? δεν είναι την ζήτηση ίδια. Ο κ. Χόβιτ. Α, όταν θα φύγουν οι Τούρκοι μάλιστα. Ίσως σε 30 χρόνια να σκέφτεστε διαφορετικά, λέει ο κ. Ματσάκης. Εγώ δεν θα κάνω σχόλια για την ιδέα του κ. Ματσάκη, αλλά χαίρομαι που τουλάχιστον για μία φορά δεν επικρίνει την, τις Βρετανικές ένοπλες δυνάμεις, αλλά κάποιες άλλες. Ίσως δεν έπρεπε να κάνω το αστείο αυτό πρόεδρε. Σύντομα, μία συγκεκριμένη ερώτηση σε κάθε έναν από τους ομιλητές. Λουκιάνοφ. Άκουσα προσεκτικά τα όσα είπατε σχετικά με, την ακαταλληλότητα του να βασίζεται κανείς σε ε, ε, θεσμούς δυτικού χαρακτήρα. Ανθρώπινα δικαιώματα στην Τσετσενία, ε, η μεταχείριση ομάδων που ενδιαφέρονται για δημοκρατικές ε, διαδικασίες. θα πω στις λεπτομέρειες, ε, ασκούνται διάφορου κριτικές διαφώνησαν κριτικέ κριτικές για αυτά τα πράγματα. Εσείς λέτε πάντοτε ότι αυτά είναι ε, ε, δυτικότροπα, αλλά μη λησμονείτε ότι αυτά τα πράγματα είναι βασισμένα στη διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κύριε Λουκιάνοφ. Γνωρίζετε τις ε, συζητήσεις για την ε, παγκοσμιότητα των ανθρώπινων δικαιωμάτων κτλ. Πώς θα γεφυρώσουμε το χάσμα που μας χωρίζει. Κύριε Μόσες, η ανάλυση σας σχετικά με τη γειτονική σχέση είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Αλλά θα το αμφισβητήσω. Αν δεχτούμε την προϋπόθεση ότι υπάρχει κάποια δυναμική αλλαγή, παγκοσμιοποίηση, τότε η εξωτερική μας πολιτική και η δική μας σχέση της Ρωσίας έχει λιγότερη σχέση με την άμεση γεωγραφική μας σχέση, αλλά με ε, χώρες που βρίσκονται και παντού αλλού. Δεν μιλήσατε για αυτό το θέμα στην παρουσίασή σας, ίσως λόγω χρόνου. Έχω την αίσθηση ότι εάν κάποια από τα θέματα αυτά, τα οποία αποτελούν προβλήματα για την εξωτερική πολιτική της Ένωσης, όπως Ιράν, όπως Ισραήλ-Παλαιστίνη. Θα μπορούσαμε ε, και για αυτά να έχουμε, να έχουμε καλύτερη σχέση με τη Ρωσία, εάν η Ρωσία ήταν διατεθειμένη να κινηθεί όπου ίσως υπάρχει και επικαλυπτόμενα συμφέροντα, αν και δεν ταυτίζονται, για αυτές τις ε, περιοχές. Και αυτό θα ήταν εξαιρετικό για τις αμοιβαίες μας σχέσεις. Μήπως μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό. Και Τέλος κύριε Κοσατσόφ, όπως η συνάδελφός μου των Πρασίνων και σχεδόν όπως, φίλος μου, όπως ο φίλος μου ο κύριος Ματσάκης, θέλω να κατανοήσω καλύτερα εάν η ιστορική συζήτηση στη Ρωσία λέει ότι η Ρωσία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και θέλει να αποτελέσει και μέλος της Λέσχης. Δεν μιλώ μόνο για τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά για την οικογένεια γενικότερα. Τι σημαίνει στην πράξη αυτό. Ποιε είναι οι άμεσε συνέπειε από αυτή την τάση. Δηλαδή τι θα κάναμε διαφορετικά μαζί ή θα κάνει η Ρωσία στο μέλλον διαφορετικά από αυτά που κάνει σήμερα. Γιατί αλλιώ μένουμε στο πολύ θεωρητικό επίπεδο. Εάν δεν συναγάγουμε κάποια συμπεράσματα για τις πρακτικές επιπτώσεις στην περίπτωση αυτή. Ευχαριστώ κύριε Χάουτο, κύριε Ζαλέσκι. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα απλό ερώτημα για τον κύριο Κοζατσόφ. Αν μπορείτε να προβλέψετε αν θα υπάρξει στρατηγική εταιρική σχέση, πρέπει να ξέρουμε κάτι σε σχέση με το τι θέλουν οι λαοί. Και κάντε μια διάκριση μεταξύ αυτών που προτιμούν την ε, μεγάλη Ρωσία από την προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σκέφτονται οι νέοι, αυτοί που είναι 20-25 χρόνων, αυτοί που θα έχουν εξουσία σε 10-15 χρόνια, τι σκέφτονται. Τους ενδιαφέρει η μεγάλη Ρωσία ή θέλουν μια μεγαλύτερη προσέγγιση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία. Χάνεται κάπου ο αντιαμερικανισμός και αντικαθίσταται από μια ευρωπαϊστική φιλοσοφία τι <clears throat> σκέφτονται οι που κάποτε σε 10-15 χρόνια θα εκπροσωπούν εδώ την ε, Ευρώπη. Ο Σάξ από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω τη μυθική μου γλώσσα. Στον κύριο Κώστατσεφ θέλω να θέσω το εξής ερώτημα. Είπατε ότι το πρόβλημα σήμερα είναι ότι δεν έχει προκύψει καμιά απόφαση αν η Ρωσία και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απλή εταίροι ή στρατηγική εταίροι. Εμείς από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε τονίσει πως βλέπουμε εμείς αυτήν τη σχέση. Ίσως είναι αυτή η διαφορά κατανόησης των αξιών που αποτελεί ένα εμπόδιο για τη σχέση μας, αλλά αναρωτιέμαι πώς σκέφτεται η Ρωσία αυτά τα θέματα. Τι θεωρείτε ότι είναι το εμπόδιο για να μπορέσουμε να καθορίσουμε τη σχέση μας ως μια απλή εταιρική σχέση ή μια στρατηγική σχέση. Τι πιστεύει η Ρωσία για όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και ο πρόεδρος, ο κύριος Χόρατσεκ από τις Πράσινους έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Στη συζήτηση που έχει γίνει έχουμε θίξει περίπου όλα τα στοιχεία του επιστητού αλλά εγώ θα ήθελα πλησιάσω την προβληματική αυτή από την άποψη ενός ατόμου που θέλει να δημιουργήσει μια οικογένεια. Είναι μια διαφορετική αντιμετώπιση της στρατηγικής εταιρική σχέσης. Τότε πρέπει να είναι κανείς προσεκτικός ακόμα και καχύποπτος. Αν δει ποιο είναι το παρελθόν των εταίρων, δεν μπορεί κανείς να ασχοληθεί μονάχα και να δει τα θετικά στοιχεία, τα στοιχεία τα οποία είναι ευάρωστα στην δυνητική σύντροφό του, να δει αν είναι ευηδής η δυνητική εταίρος του και να δει μονάχα αν έχει πρίκα και εδώ εννοώ φυσικούς πόρους. Θα πρέπει κανείς να σκεφτεί και το μέλλον και να χρησιμοποιήσει την κεκτημένη εμπειρία του παρελθόντος για να προβλέψει καλύτερα το μέλλον. Και όταν λέω για μας εννοώ για αυτούς από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη που προέρχονται από την κεντρική και ευρωπαϊκή, ανατολική Ευρώπη και οι οποίοι έχουν ακόμα την ανάμνηση <clears throat> της στρατηγικής συμμαχίας με την Ρωσία στα πλαίσια της Σοβιετικής Ένωσης και του συστήματος αυτού. Η συνθήκη της Ρώμης, όπως μας υπενθύμησε ο πρόεδρος Μπαρόσο όταν πρέπει να αντιμετωπίζεται από τον πρόεδρο τότε Πουτίν, ο οποίος ήταν πρώην πράκτορ της ΚΑΓΕΜΠΕ, αυτό δείχνει μια απόκληση και μια διαφορά μεταξύ των δύο πλευρών, διότι τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν παραβιαστεί στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Όλο αυτό μας ε, κάνει να σκεφτούμε και για θέματα όπως η αντιμετώπιση του και που είναι στη φυλακή, την αντιμετώπιση του Γιούκος για τη δολοφονία δημοσιογράφων. Όλα αυτά συγκροτούν μια προβληματική την οποία δεν μπορούμε να την παραγνωρίσουμε. Και όταν ακούω από τον κύριο Σφάτσεμπερκ, τον Υπουργό Εξωτερικών της ε, ε Τσεχίας, ότι όταν θίτουμε ορισμένα προβλήματα στη Ρωσία ε, Μα απαντά ο Υπουργό Εξωτερικών τη Ρωσία, ο κ. Λαυρόσκι, Μα εσεί είσαστε από την Ανατολική Ευρώπη και αυτό δεν είναι μόνο ένα γεωγραφικό προδιορισμό. Όλα αυτά δεν αποτελούν για μένα μία ευσταθή βάση για την δημιουργία μια οικογένεια και μια εταιρική σχέση, και πάλι όχι επειδή βρίσκω μια όμορφη κοπέλα. Δεν σημαίνει αυτό μια όμορφη και πλούσια κοπέλα ότι αυτό αρκεί για να φτιάξω μια οικογένεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Χόρατσακ. Ο κύριος Βιλαβίσκη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι ευχαριστώ θερμά και τους δύο εμπειρογνώμονες, τον κύριο Λουκιάνοφ και τον κύριο Μόησος, για την ακριβέστατη, λεπτομερέστατη, ενδελεχέστατη παρουσίαση των προβλημάτων και τη θαραλέα παρουσίασή τους. Έχω κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά αυτά που είπατε, αλλά ήταν μια άριστη εισαγωγή. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον πρώην συνάδελφο του Συμβουλίου της Ευρώπης, τον κ. Κωνσταντίν Κασάτσεφ, που παρουσίασε το δίλημα για τη Ρωσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση σωστά. Δηλαδή μιλάω για τι αμοιβέ μας σχέσει. Εντό της νέας γενιάς, για να το πω ήπια, άντε στα επόμενα χρόνια θα πρέπει να γίνουν αρκετέ επιλογές. Και με βάση αυτές τις επιλογές θα δούμε κατά πόσο θα γίνουμε μια κοινή ευρωπαϊκή οικογένεια ανεξάρτητα από την πολιτική μορφή που θα έχει ή θα είμαστε απόμακροι συνεργάτες με τη Ρωσία. Δεν θα θέσω κάποια ερωτήματα, διότι τα ερωτήματα που ετέθησαν από τον κύριο Ρόιτσε και τον κύριο Σβόμποντα για τις σχέσεις ε, γειτονίας με τους γείτονες της Ρωσίας είναι σημαντικότατες ερωτήσεις. Έχω δύο επιφυλάξεις όσον αφορά αυτά που είπατε. Δεν συμφωνώ με τον κύριο Λουκιάνοφ σχετικά με το όραμα παρουσίας για τις προπτικές. Υπάρχει κάποιο όραμα, είναι προφανές. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε παράμερα. Εντός των επομένων 25 ετών, φεριπίν, θα έχουμε μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία αναδιαθρώσεως των ενεργειακών δομών και οι χώρες που έχουν δικούς τους ενεργειακούς πόρους θα πρέπει γρήγορα να βρουν διαφορετικές οικονομικές δομές. Όπως βλέπουμε τα πράγματα σήμερα, πιστεύω ότι η Ρωσία δεν θα έχει επιλογή και είπα δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα σχετικά και δεν πρόκειται να κάνουν πολλά σχετικά. Η στενή συνεργασία με την Ινδία και την Κίνα είναι κάτι αμφίβολο και πολύ δύσκολο, κυρίως όσον αφορά τους πολιτικούς στόχους που επιδιώκουν οι δύο αυτές χώρες και κυρίως αλάβουμε υπόψη τον κινέζικο εθνικισμό. Άρα είμαστε καταδικασμένοι να δούμε μαζί. Σας χρειαζόμαστε σήμερα ιδιαίτερο όσον αφορά τον εφοδιασμό σε ενέργεια και η Ρωσία θα χρειαστεί εμάς και στενή συνεργασία μαζί μας σχετικά με τις επενδύσεις, με την τεχνολογία, διαχείριση επιχειρήσεων και ελεύθερη αγορά ούτως ώστε να μπορέσει η Ρωσία να αλλάξει τις οικονομικές της ε, δομές. Και αυτό είναι ένα αναπόφευκτο σαν πρόκληση. Θα πρέπει να δεχτούμε αυτή την πρόκληση μαζί. Διότι για μας στις παγκόσμιες εξελίξεις αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντικά. Και είμαστε αναγκασμένοι να συμβιώσουμε. Και δεύτερο σχόλιο που απευθύνω προς τον κύριο Κωνσταντίν Κοζάτσεφ. Το τεστ, η δοκιμή που θα γίνει τα επόμενα χρόνια και θα διαπιστώσουμε αν θα είμαστε στενοί εταίροι ή ανταγωνιστές θα είναι το εξής. Θα είναι το θέμα της ενέργειας και της ενεργειακής ε, πολιτικής. Η εξελίξη στον τομέα της ενέργειας, η ανάπτυξη της σχετικής τεχνολογίας. Νομίζω ότι η Ρωσία δεν θέλει να παραδεχτεί λόγω των δικών της συμφερόντων ότι εμείς εδώ στην Ευρώπη κυρίως βάσει των εμπειριών των τελευταίων μηνών, θα πρέπει να βρούμε διαφορετικές πηγές ενέργειας και διάφορες μεθόδους για τη χρήση της ενέργειας. Θα πρέπει να αλλάξουμε λοιπόν τις μορφές ενέργειας που χρησιμοποιούμε, για να το πω απλά. Θα πρέπει να περιμένουμε λοιπόν συνεργασία, καλή βούληση σε πλευράς της Ρωσίας. Και εδώ είναι σοβαρότατη δοκιμή αυτή, διότι η ασφάλεια της Υπήρου μας εξαρτάται από την επίλυση αυτών των σημαντικών προβλημάτων των σχετικών με την ενέργεια. Θα είναι μια δοκιμή που θα δοκιμάσει την καλή μας βούληση και ελπίζω να έχουμε τελικά επικοδομητική συνεργασία με το ΣΥΚΙ ε, Ομοσπονδία. Ξεπεράσαμε τα χρονικά όρια γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα, λέει ο Πρόεδρος. Τώρα είναι η ώρα, έστω και καθυστερημένα, να απαντήσει το πάνελ στις ερωτήσεις και τα σχόλια. Θα ακολουθήσουμε αντίστροφη σειρά από ό,τι όταν αρχίσαμε, ξεκινώντας από τον Κωνσταντίν Κοζατσόφ. Επιτρέψτε μου να μιλήσω ρωσικά, λέει ο κ. Κοζατσόφ, για να προωθήσω κι άλλη μια γλώσσα στη συζήτηση. Στο κανάλι 23 θα ακούσετε ρωσικά, λέει ο Πρόεδρος, 23. Σας ευχαριστώ. Στο 2 θα ακούσετε, τα αγγλικά. Λοιπόν, έχω δύο σχόλια για την οικονομική κρίση και τις συνέπειες που έχει η οικονομική κρίση για, σε σχέση με τη διεθνή πολιτική που ακολουθεί η Ρωσική Ομοσπονδία. Το πρώτο πράγμα που έχω να πω σχετικά με αυτό είναι ότι είμαστε μέσα στην κρίση και μας επηρεάζει η κρίση και δραματικά και οι συνέπειες της κρίσης αυτής δεν διαφέρουν στη Ρωσία σε σχέση, σε σύγκριση με τις άλλες χώρες και τις χώρες Ευρωπαϊκής Ενώσεως και όταν ακούω διάφορα πράγματα που λέγονται, δηλαδή τι μπορεί να κάνει για τη Ρωσία Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαι ευγνώμων για αυτά που λέγονται, αλλά έχω την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρειαστεί βοήθεια και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα χρειαστούν κάποια βοήθεια κατεπηγόντως. Η Ιρλανδία και η Λετωνία χρειάζονται βοήθεια σε αυτή τη φάση και θα χρειαστούν και άλλες χώρες στον κατάλογο που περιμένουν για βοήθεια και οι γειτονικές μας χώρες, η Ουκρανία Φερρυπίν, θα αισθανθεί πιο επιβλαβείς συνέπειες από την οικονομική κρίση από τη Ρωσία και βλέπω να υπάρχει στενή σχέση με τις συζητήσεις για πολιτικά συστήματα και δημοκρατία. Πιστεύω ότι το ουκρανικό πολιτικό σύστημα με όλες τις δημοκρατικές προσδοκίες δεν είναι βιώσιμο σύστημα στα πλαίσια αυτών των συνθήκων της χρηματοπιστωτικής κρίσεως και η Ρωσία ανησυχεί τα μάλα για αυτές τις ε, εξελίξεις. Σίγουρα πιστεύω ότι στην εξωτερική μας ε, πολιτική που επηρεάζεται από την οικονομική κρίση ε, δεν θα γίνει πιο επιθετική. Δεν το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την οικονομική κρίση όλοι μαζί. Και από αυτή την έποψη για μας η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο βασικός στρατηγικός και υπογραμμίζω στρατηγικός ε, εταίρος όσον αφορά την οικονομία. Και όταν τίθεται το θέμα που έθεσε ο κ. Γκάλερ γιατί η Ρωσία δεν επιτρέπει τους ξένους επενδυτές σε στατηγικούς τομείς δραστηριοτήτων υπάρχουν δύο απαντήσεις που μπορούν να δοθούν. Πρώτα απ' όλα θα έπρεπε να είναι αμφίδρομη αυτή η σχέση και μπορώ να σας δώσω πολλά παραδείγματα περιορισμών που αντιμετωπίζουν οι Ρώσοι. Ρωσικά κεφάλαια και Ρώσοι επενδυτέ δεν μπορούν να επενδύσουν σε στρατηγικού τομεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ξέρετε αυτά τα παραδείγματα, δεν πρόκειται να αναφερθώ λεπτομερώ σε αυτού του τομεί. υπάρχει άλλο πρόβλημα. Τι περιμένουν οι καταναλωτέ. Πολλοί ευρωπαϊκέ επιχειρήσει τείνουν να εκμεταλλεύονται την. περιουσία ε, της Ρωσίας και είδαμε τη σύγκρουση BP και TNK στη Ρωσία. Όπως και να τα δει κανείς τα πράγματα, είδαμε ότι οι Βρετανοί επενδυτές σε αυτή την περίπτωση προσπάθησαν να εμποδίσουν την κοινοπραξία που πήγε να δημιουργηθεί για να χρησιμοποιηθούν οι νέοι πετρελαϊκοί πόροι υπέρ της χρήσης υφισταμένων ε, πόρων, κάτι που δεν μπορούσαν να δεχθούν οι ρωσικές συνιστώσεις της κοινοπραξίας. Δεν θα πει σε λεπτομέρειες, δεν υπάρχει χρόνος. Αυτά ήθελα να πω εν είδη εισαγωγής. Όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Ρωσίας, κατά πόσο μπορεί η Ρωσία τελικά να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώση και πώς το βλέπει η κοινή γνώμη στη Ρωσία και ποια είναι η άποψη της νεολαίας. Δυστυχώς, και εκφράζω προσωπική άποψη που μοιράζομαι μαζί σας, δυστυχώς η ιδέα του ε, δεν είναι τόσο δημοφιλής ιδέα και μειώνεται η, το πόσο ελκυστική είναι αυτή η ιδέα. Γιατί το λέω αυτό. Του να συμμετέχει, να γίνει μέλος της, Ευρωπαϊκή, της Ευρωπαϊκής ως η Ρωσία. Δεν βλέπουμε εμείς την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν κοινότητα των αξιών, σαν Ρώση, όπως την αναφέρετε εσείς. Σε αρκετές περιπτώσεις βλέπουμε διπλά μέτρα και διπλά σταθμά από πλευρά Ευρωπαϊκή Ενώσεως. Αυτό το μήνυμα περνάει. Μα κατηγορείτε για την κατάσταση στη Γεωργία, αλλά σα υπενθυμίσω εγώ το βομβαρδισμό του Κωσυφοπεδίου, όταν οι δυνάμει του ΝΑΤΟ όχι μόνο βομβάρδισαν στατιωτικούς στόχους, αλλά βομβάρδισαν και την πρωτεύουσα της Σερβίας, το Βελιγράδι. Εμείς δεν βομβαρδίσαμε ποτέ την Τυφλίδα, την πρωτεύουσα της Γεωργίας, αλλά το ΝΑΤΟ το έκανε αυτό στο Βελιγράδι. Και εδώ χωρίζουν οι δρόμοι μας όσον αφορά τις αξίες. Μία ενωμένη Ευρώπη ζητά από τη Ρωσία να λύσει το πρόβλημα των προβλημάτων των μειονοτήτων στη Ρωσία που αρκετές χιλιάδες δεν είχαν καθεστώς ε, υπηκότητας ρωσικής τουρκόφωνων πολιτών και αυτό θεωρείται απάνθρωπο. Αν σας δώσετε και άλλα παραδείγματα, Λετωνία και αλλού, υπάρχουν παρόμοια προβλήματα. Και μπορούμε να συνεχίσουμε αυτά τα παραδείγματα. Αν μιλάμε για την νεολαία, έχουμε μία τάση που χαρακτηρίζει τη ρωσική νεολαία όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα θυμόσαστε τα γεγονότα στο κέντρο του Ταλίν, στην πρωτεύουσα της ε, Εστονίας. Πολλοί νέοι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις και στη Ρωσική Ομοσπονδία δεν σπάσαν τίποτα, δεν έκαναν τίποτα κακό, πήγαν να διαδηλώσουν οι νέοι. Και μεταξύ αυτών ήταν και ο πρόεδρος της Επιτροπής Υποθέσεων ε, Νεολαίας. Και οι αρχές της ε, Εστονίας τον έβαλαν σε μαύρο κατάλογο και δεν μπορεί να μπει σε καμία χώρα της ε, Σέγγεν. Δεν έκλεψε κανέναν, δεν κατέστρεψε τίποτα είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής για θέματα νεολαίας και είναι ένας άνθρωπος που έχει κάποιο κύρος και είναι σε μαύρη λίστα. Και δεν νομίζω ότι αυτό προβάλλει το πόσο δημοφιλής είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για τους νέους στη Ρωσία. Τρίτον, σε ποιο βαθμό η Ρωσία αντιμετωπίζει ισότιμα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εξακολουθεί να ξεχωρίζει κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ρωσία όσον αφορά την αντιμετώπιση της λόγω γεωγραφικής σχέσης, λόγω ιστορικών σχέσεων κλπ. Ο κ. Πάσκουα το έθεσε το θέμα. Δεν ξεχωρίζουμε τις χώρες Ανατολικής Ευρώπης από τις άλλες χώρες. Δεν προσπαθούμε να διατηρήσουμε την παλιά σφαίρα επιρροής Σοβιετικής Ένωσης. Καταλαβαίνουμε ότι προχωράει η Ευρωπή προχωράει ο κόσμος και εμείς προσαρμοζόμαστε δεόντως. Όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις με κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, πράγματι καμιά φορά αυτές οι διμερείς σχέσεις ε, μερικές διμερείς σχέσεις είναι πιο καρποφόρες από ότι οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν σύνολο. Ας πούμε για άρση των προξενικών θεωρήσεων. Θα θέλαμε να αρθούν οι ε, ε, θεωρήσεις με όλες τις χώρες, για όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Μας είπαν ότι αυτό είναι ανέφικτο. Έπρεπε να βρούμε λύσεις με Γερμανία, με Γαλλία, με Ιταλία και επελήφθη το πρόβλημα. Ήταν αρκετά εύκολα τα πράγματα. Αν θέλουμε να προχωρήσει και να λυθούν τα προβλήματα εν γέννη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, Εάν βελτιωθεί γενικά αυτό το πρόβλημα με όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι καλύτερη λύση και ελπίζω κάποια μέρα δεν θα υπάρχουν περιορισμοί ε, προξενικών θεωρήσεων. Τώρα για τις γειτονικές χώρες, Λευκορωσία, Κυργιζιγιστάν, ε, εγώ συμφωνώ ότι η Ρωσία δεν θα πρέπει να έχει κάποια πλεονεκτήματα και να διεκδικεί κάποια δικαιώματα όσον αφορά τα εδάφη αυτών των χωρών. Τούτων λεχθέντων όμως εγώ δεν συμφωνώ με την ιδέα ότι εμείς δεν θα πρέπει να έχουμε κάποια ωφέλη ε, ε, στη σχέση με αυτές τις χώρες γιατί είναι οι άμεσοι γειτονές μας οι πιο κοντινοί ε, γειτονές μας. Να έχει μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση πολιτική γειτονία. Σε αυτό τον όρο το χρησιμοποιούμε επί 15 δεν χρησιμοποιούμε πια τον όρο πολιτική γειτονία και κοντινοί γείτονε, πολιτική γειτονία. Λέμε οι κοντινοί μα γείτονε, οι γείτονέ μα. Δεν χρησιμοποιούμε πια αυτόν τον όρο πολιτική γειτονία. Συμφωνώ με τον κύριο Σβόποντα. Θέλουμε να έχουμε πολύ καλέ σχέσει ε, με τους γειτονές μας. Πέμπτο σημείο, η Γεωργία. Νομίζω ότι αξίζει κανένα δίλεπτο να επεκταθούμε επί της Γεωργίας, διότι υπόθηκαν κάποια πράγματα. Είπατε ότι η Ρωσία κατέκτησε, κατέχει, ήταν εισβολές κλπ. Πρώτα απ' όλα σας απευθύνω μια έκκληση. Παρακαλώ, καταλάβετε το, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταλάβετε λοιπόν ότι η Γεωργία δεν υπήρχε, δεν υπήρχε σαν κυρίαρχο κράτος όταν διακήρυξε την ανεξαρτησία της, αυτή ήταν μια διακήρυξη de jure που έπρεπε να αποδειχτεί de facto. Και η Ρωσία επί 18 χρόνια προσέφερε τη δυνατότητα στη Γεωργία να είναι κυρίαρχο κράτος, να δημιουργηθεί σαν κυρίαρχο κράτος. Διότι υπήρχαν προβλήματα εθνοτήτων στη Γεωργία που έπρεπε να επιληθούν. Ξεκινήσαν τα προβλήματα δεκαετία του 80, μετά συνεχιστήκαν τη δεκαετία του 90 και, συνεχίστηκαν και στον 21ο αιώνα. Προσπάθησε να χρησιμοποιήσει βία η Γεωργία και να υποχρεώσει τους Απχάζους και τους κατοίκους της Νότιας Οσετίας να συνεπάρξουν. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί με τη βία, μπορεί να γίνει με αμοιβαία αποφελή τρόπο. Παραδείγματο χάρη έχουμε Σερβία, Κωσυφοπέδιο. Όλοι είναι έτοιμοι εκεί να αποδεχτούν την πραγματικότητα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει, είναι αντανάκλαση αυτής της καταστάσεως και στη Γεωργία. Και θέλω να το επαναλάβω. Λυπούμε πολύ ότι η ίδια ακριβώς κατάσταση επικρατεί στην Απχασία και Νότια Οσετία, συγγνώμη, στη Γεωργία. Και όταν μιλάμε για τις δράσεις των Ρώσων, Εκεί δεν μιλάμε για δράση, αλλά αντίδραση. Ήταν αντίδραση στις δολοφονίες των Ρώσων πολιτών και εκείνων που προσπαθούσαν να επιβάλλουν την ειρήνη. Και όταν κατηγορείται σήμερα η Ρωσία ότι πολεμά, χρησιμοποιεί όπλα για να προασπιστεί την ασφάλεια των πολιτών της, αυτό ακούγεται πάρα πολύ τρομακτικό, αλλά δεν αληθεύει. Αν οι πολίτες όμως της Ρωσίας δολοφονηθούν, αν σκοτωθούν, εμείς θα τους υπερασπιστούμε και κάθε ευρωπαϊκή χώρα θα ακολουθούσε ακριβώς την ίδια αντιμετώπιση. Είναι μια υποθετική κατάσταση αυτή βεβαίως και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να τη συζητήσουμε και να μπούμε σε βάθος. Και το τελευταίο θέμα το οποίο θα ήθελα να θίξω είναι η συνεργασία στον ενεργειακό τομέα, συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, και Ρωσίας και πώς μπορεί να δηλαδή διάφορες μορφές αυτή η συνεργασία. Λοιπόν, πώς θα πετύχει αυτή η ενεργειακή συνεργασία. Πρέπει να το εξετάσουμε το θέμα. Δείτε τι έχει γίνει κατά το παρελθόν. Είδαμε τι γινόταν με τη διοχέτευση πετρελαίου μέσω της Βαλτικής προς την Ευρώπη. Υπάρχει ένα εναλλακτικό σύστημα. Στις αρχές του δεκαετίας του 90 οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και των Βαλτικών χωρών δεν ήταν και οι καλύτερες. Και η διέλευση ε, τώρα ακολουθεί, η διέλευση ενέργειας ακολουθεί εναλλακτικό δρόμο. Μιλάμε για το North Stream και το South Stream και έχουν γίνει σημαντικοί ε, διάβλοι διότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην Ουκρανία. Και έχουμε αποτύχει θα έλεγα όλοι μας διότι θα προτιμούσαμε να μην κατασκευάζουμε νέους αγωγούς και να χρησιμοποιήσουμε τους υπάρχοντες αγωγούς. Διότι η δίωδος μέσω της Ουκρανίας είναι η συντομότερη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όμως αντιμετωπίζουμε σήμερα πρόκληση. Εστιαστήκαμε στις ευθύνες ε, της Ρωσίας, που είναι ο προμηθευτής της ενέργειας. Και εθελοτυφλήσαμε όσον αφορά τη χώρα διέλευσης που είναι η Ουκρανία. Η Ουκρανία προσπάθησε να καταχραστεί την φτής σαν χώρα διέλευσης. Και τώρα προσπαθούμε να την υπερκεράσουμε. Επενδύουμε χρήματα για να βρούμε εναλλακτικούς αγωγούς και από βόρεια και από νότια. Τεράστια ποσά δίνουμε, καταβάλουμε. Δεν θα κατασκευάσουμε λοιπόν αγωγούς και μετά θα τους αποκόψουμε. Αυτό δεν θα τέριαζε με τα βασικά μας οικονομικά συμφέροντα. Βασικό μας συμφέρον είναι να έχουμε πάρα πολύ ευρεία ε, και στενή συνεργασία στον ενεργειακό τομέα με την Ευρώπη. Αν είναι επιτυχές το πρόγραμμα Ναμπούκο και σχετικά άλλα προγράμματα, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, δεν θα δημιουργήσει η Ρωσία κανένα πρόβλημα. Σίγουρα ε, επικρατεί οικονομική λογική όσον αφορά την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων. Όταν η, η δική μας αγωγή στο Nord Stream και στο South Stream αποκοπούν για πολιτικούς λόγους από τη Σουηδία, τις Βαλτικές χώρες και λοιπά, είμαστε κατά αυτής της αντιμετωπίσεως. Εκατακλείδη, η Ρωσία έκανε κάποιες επιλογές. Για μας η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας στατηγικός εταίρος και οι συνομιλίε που μπαίνουν στον τρίτο γύρο του, ξεκινάει ο τρίτο γύρο των συνομιλιών αύριο, οι συνομιλίε αυτέ λοιπόν θα είναι σημαντικέ για μα. Θα προσφέρουμε στου εταίρου μα στην Ευρώπη του όρου για τη στρατηγική αυτή συνεργασία και θα αποφασίσετε εσεί. Ευχαριστώ για αυτέ τι δηλώσει, για καλέ προθέσει λέει ο Προεδρο. Θα δοκιμάσουμε αν οι προθέσει αυτέ θα αποκρίνουν στην πραγματικότητα. Ο, ο κ. Μόσος έχει το λόγο τώρα. Thank you, Mr. Chairman, as we're really running behind Αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε καθυστερήσει. Θα είμαι σύντομος. Θα απαντήσω σε ορισμένε από τι ερωτήσει που τέθηκαν. Συμφωνώ με την δήλωση που λέει ότι πρέπει να κάνουμε μια διαφοροποίηση μεταξύ χωρών και να δούμε την κάθε χώρα και τις δικές της ιδιότητες ικανότητες. Υπάρχει όμως ένας τρόπος να συμπεριλάβουμε και μια γενίκευση. Κάθε χώρα που είναι μέλος της κοινοπολιτείας ανεξάρτητων κρατών κάνει τη δική της προσπάθεια. Ακόμα και αν εν μέρη εξαιρέσουμε την Ουκρανία η οποία κάνει τα δικά της ακροβατικά προς τα μέσα. Οι υπόλοιπες χώρες προσπαθούν να κρατήσουν κάποιες ισορροπίες μεταξύ σε, ε, μεταξύ της Ρωσίας και της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις περιπτώσεις των χωρών του Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας <coughs> προσπαθούν να ισορροπήσουν μεταξύ Ρωσίας, Κίνας, ε, Δύσης, ορισμένων τοπικών ας πούμε δυνάμεων όπως της Τουρκίας δεν θα μπορέσω να επεκταθώ περισσότερο όπως θα ήθελα αλλά αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τις ε, γεωγραφικά δυτικές χώρες της κοινοπολιτείας το γεγονός ότι μέσα στα 15, 16, 17 χρόνια έχουν αρχίσει και απομακρύνονται από την Ρωσία και η επιρροή, σε αυτές έχει, ε, επιρροή της Ρωσίας σε αυτές έχει μειωθεί και η ελκυστικότητα της Ευρώπης έχει αυξηθεί σε όλες αυτές τις χώρες και στο Αζερβαϊτζάν. Για μένα αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Το γεγονός ότι και οι έξι χώρες Ουκρανία, Λευκορωσία, Μολδαβία και τρεις χώρες του Καυκάσου συμμετέχουν από την αρχή στην πολιτική γειτονία και τώρα μπαίνουν και στην ε, εταιρική σχέση με την Ανατολή, στην οποία δεν συμμετέχει δομικά η Ρωσία. Αυτό είναι σημαντικό σημάδι μιας ποιοτικής αλλαγής. Θα υπάρξει και ένας νέος γύρος αλληλεγγύης αδύναμος μεν, αλλά με επίκεντρο την Ευρώπη και όπου η Ρωσία δεν θα αποτελεί μέλος. Και αυτό βέβαια είναι το αποτέλεσμα των τελευταίων εξελίξεων, των 20 ετών δηλαδή. Δεν θα ε, αναφερθώ περισσότερο σε αυτό το θέμα τώρα. Σφαίρα επιρροής. Ίσως η ερώτηση τέθηκε προς εμένα επειδή εγώ χρησιμοποίησα τον όρο αυτό αλλά δεν είμαι και ο πλέον κατάλληλος για να απαντήσω στην ερώτηση αυτή από όσους συμμετέχουν στο πάνελ, διότι εργάζομαι, εργάζομαι σε ερευνητικό ίδρυμα που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Φιλανδικού Κοινοβουλίου και όχι της Ρωσικής Δούμας. Εγώ δεν συμφωνώ με τη λογική που υπαγορεύει τον όρο αυτό, αλλά τούτων λεχθέντων θα πω επίσης ότι είναι περίπλοκο το θέμα. Εάν η Ρωσία, η Μόσχα ή τέλο πάντων κάποιοι στην Μόσχα ε, ε, ε, μιλούν για το δόγμα της σφαίρας προνομιούχων συμφερόντων. Εάν βέβαια υπάρχει ο ισχυρισμό αυτός, η αξίωση αυτή, εάν αυτή γίνει δεκτή σε ορισμένες, αναγνωριστή σε ορισμένες γωνιές του δυτικού κόσμου. Επειδή ορισμένοι στην Δύση θεωρούν καλύτερα να μην ανακατεύονται πολύ προς τα δυτικά, προς τα ανατολικά μάλλον των ε, ανατολικών συνόρων της Ένωσης, θα ε, επιληφθεί η Ρωσία. Και πάλι τον 2008 θα μπορούσε να έχει αποτελέσει ένα είδος κατόφλι η ευρωπαϊκές φιλοδοξίες σχετικά με την Ουκρανία δεν έγιναν, δεν υλοποιήθηκαν και δεν μιλώ για αυτές του ΝΑΤΟ, για Ουκρανία-Γεωργία, γιατί εκεί η απόφαση είχε κάποια λογική. Είναι πολύ δύσκολο να προωθηθεί η προοπτική του ΝΑΤΟ για τις δύο χώρες αυτές σε χώρες όπου η μία τουλάχιστον ε, η πλειοψηφία εκεί είναι αντίθετη και η άλλη έχει προβλήματα στα σύνορά της δεν μιλώ εδώ για το θέμα λοιπόν τη ενδεχομένη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ, αλλά τη προοπτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρχε στην Ουκρανία πλειοψηφία υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής για χρόνια. Ποτέ στα ανοιχτά. Ποτέ δεν ανοίχτηκε ρητά και αδιαμφισβήτητα. Και αν νομίζετε ότι το γεγονός αυτό δεν ενθάρρυνε τους υποστηρικτές της σφαίρας επιρροής της σχετικής νοοτροπίας στη Ρωσία, τότε ε, κάνετε κάποιο λάθο. διότι όντως τους ενεθάρρυνε ε, το γεγονό ε, ότι το όριο ανάμεσα στον ενοποιημένο χώρο του ΝΑΤΟ και στο μη ενοποιημένο χώρο, ρωσικό χώρο, δεν επαφείται μοναχά στο τι σκέφτονται ορισμένοι στη Ρωσία, αλλά τι σκέφτονται και άλλοι αλλού. Και αναλυτικά θα ήταν εσφαλμένο να ρηχθεί το βάρος της ευθύνης μονάχα στη ρωσική πλευρά. Το πρόβλημα είναι ότι οι σχετικές ρητορίες της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής αλλά και η σχετική νοοτροπία είναι ε, εκπληκτικά διαφανής σε πολλά θέματα. Οι Ρώσοι λένε πραγματικά αυτό που πιστεύουν. Ακούσαμε εδώ για ένα στοιχείο του δόγματος Πούτιν Μετβιέντεφ πάλι σχετικά με την δηλωμένη πρόθεση της Ρωσίας να χρησιμοποιήσει και βία για να προστατεύσει τους Ρώσους πολίτες στο εξωτερικό. Αυτό όμως δεν είναι μέρος μόνο του δόγματος Πούτιν με τη Ρετεφή. Υπήρχε πάντοτε. Διαβάστε τα έγγραφα της δεκαετίας του 90. Η διαφορά είναι ότι στη δεκαετία του 90 η ε, Ρωσία δεν είχε τη δύναμη να υλοποιήσει τα όσα έλεγε. Αλλά το 2008 το έκανε και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να πάει στη Μόσχα και να πει μα, καλά αυτά που λέγατε τα εννοούσατε και πραγματικά και χρειάστηκε ο πρόεδρος να πάει δηλαδή να πάει και δεύτερη φορά στην Μόσχα και για να κάνει το ίδιο ερώτημα και να το απαντήσουν ναι πραγματικά τα εννοούσαμε αυτά που λέγαμε πρέπει να αντιληφθείτε τώρα την διαφάνεια και την ειλικρίνεια ορισμένων από όσα λέει η Μόσχα. Και ίσως πρέπει να την ευχαριστούμε τη Μόσχα που ε, είναι ειλικρινής. Όπως γνωρίζουμε από την κλασική διπλωματία, κάθε χώρα χρησιμοποιεί το περιθώριο ελιγμών που διαθέτει. Και αυτό είναι περίπλοκο το θέμα. Ορισμένοι στην Μόσχα απεφάσισαν ότι στην παρούσα ιστορική στιγμή το περιθώριο ελιγμών που διέθετε τους επέτρεπε να αναλάβουν ορισμένες δράσεις. Και η ανάλυση τους αυτή ήταν σωστή εν τέλει, για να το πω ομά. Τώρα, για τον υπεριαλισμό. Δεν μ' αρέσει η χρήση του όρου «Ιμπεριαλισμός». Υπάρχει και ίσως μια διαφορά ερμηνείας. Εγώ τον υπεριαλισμό τον βλέπω ιστορικά. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία άρχισε με τον «Ιμπεριαλισμό» μεταφέροντας και τα φώτα της παιδείας και συνέχισαν και οι υπόλοιποι. Αυτά που κάνει η Ρωσία τώρα δεν είναι «Ιμπεριαλισμός» είναι κατανοητή πολιτική μιας ισχυρής δύναμης η οποία θέλει να έχει πελατειακές σχέσεις με άλλες χώρες. Η διαφορά και πάλι είναι ότι αυτό το κάνει χρειάστηκε μισή γενιά, χρειάστηκαν 15 χρόνια ανάπτυξη των εσωτερικών πολιτικών στην ε, Ρωσία πριν αποκρισταλωθεί αυτή η πολιτική. Σήμερα, αντίθετα από ότι πριν από 15 χρόνια, οι Ρώσοι δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για τις επιπτώσεις που έχουν ορισμένες δράσεις τους στον τομέα της ενέργειας στην οικονομία της Ουκρανίας. Πριν από 15 χρόνια θα ενδιαφέρονταν για τις επιπτώσεις αυτές, διότι υπήρχε ακόμα ιδέα ότι αυτή η αποσύνθεση της ε, πρώην Σοβιετικής Ένωσης ήταν ε, προσωρινό φαινόμενο και ότι θα επανέρχονταν ε, στους ε, κόλπους της οικογένειας κατά κάποιο τρόπο. Όταν μιλώ για υπεριαλισμό, γιατί αυτό δεν έγινε εν τέλει, δεν εννοώ ότι χάνεται κάτι και αντικαθιστάται από κάτι άλλο. Ορισμένες δράσεις και ορισμένοι στόχοι θα επιδιωχθούν κυρίως εξαναγκασμού και όχι δια της πυθούς. Αυτά χρειάζεται όμως και κάποια ανάλυση. Και εν τέλει, πράγματι δεν είχα χρόνο να αναφερθώ σε όλες τις άλλες περιοχές όπου αναπτύσσεται ρωσική εξωτερική πολιτική. Απαντώ στον κύριο Χάουιτ, θα ήταν καλό πράγματι εάν η Ρωσία συμμετείχε περισσότερο στην προσπάθεια να επιληθεί το πρόβλημα του Ιράν και η κρίση στην Μέση Ανατολή δεν είμαι ειδικό για αυτή την περιοχή του κόσμου, αλλά η ερμηνεία που δίνω εγώ είναι ότι η ρωσική πολιτική στις περιοχές αυτές ε, είναι ε, σε αντιστοιχεία με την αμερικανική πολιτική και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Ευχαριστώ κύριε Μόσες και περνάω στον κύριο Κιάνιοφ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ετέθηκαν ερωτήματα για την ε, μελλοντική δομή ασφαλείας στην Ευρώπη και ο κύριος Κοσάτσιος, τα ξέρει πολύ καλύτερα από μένα, αλλά αυτά τα οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν λειτουργεί ο ΟΑΣΕ όπως είχε σχεδιαστεί να λειτουργήσει πριν από 30 χρόνια. Θα πρέπει να επανέλθει εφόλης της κλίμακος ο ΟΑΣΕ με όλα τα καλάθια που είχε σε επίπεδο διαπραγματεύσεων στην αρχή τα θέματα ασφάλειας, τα θέματα οικονομίας και τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βρισκόμαστε τώρα σε μια κατάσταση όπου η πραγματική δραστηριότητα του ΟΑΣΕ είναι απλώς η παρακολούθηση των εκλογών. Σημαντικό θέμα, μεν, αλλά δεν αξίζει να υπάρχει ο ΟΑΣΕ μόνο και μόνο για να παρακολουθεί εκλογικές διαδικασίες. Πριν από δύο χρόνια η Ρωσία προσπάθησε να συζητήσει τα θέματα των ε, συμβατικών όπλων στην Ευρώπη και απέτυχε μέσα στα πλαίσια του ΟΑΣΕ. Αυτό το οποίο θέλει ο Μεντιεβέντιεφ είναι να αναζωογονηθούν οι συμφωνίες του Ελσίνκη. Δεν ξέρω αν αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό ή όχι, αλλά πρέπει να δούμε την πολυπλοκότητα της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας. Όταν έρχομαι στο ερώτημά σας για μια συνθήκη η οποία δεν περιέχει μια ρυθμιστική βάση. Προφανώς χρειαζόμαστε μια σαφής, σαφή ρύθμιση στα θέματα αυτά. Αυτό όμως το οποίο με ανησυχεί είναι ότι αν προσπαθήσουμε να τα συνδέσουμε όλα και να τα βάλουμε όλα μέσα σε ένα έγγραφο και να είναι όλα αλληλένδετα μεταξύ τους, δεν θα πετύχουμε το στόχο μας. Γιατί υπάρχουν τομείς όπου η συνεργασία μπορεί να ανθίσει και εκεί χρειαζόμαστε περισσότερες λεπτομερέστερες ρυθμίσεις. Σε άλλους τομείς είναι πρόωρο να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Το θέμα είναι λοιπόν ποιες περιοχές της αλληλεπίδρασής μας είναι οι περιοχές αυτές οι οποίες έχουν φτάσει αρκετό στάδιο οριμότητος για να περάσουμε στο επόμενο βήμα και εν μέρη η, τα στοιχεία που έχουμε στην τωρινή μας συμφωνία μπορεί να είναι αρκετά. Για την επιρροή στην ε, Ανατολική Ευρώπη, όπως είπε ο κ. θα ήταν κάπως ανόητο να περιμένουμε χώρες που είναι μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επανέλθουν στη ρωσική σφαίρα επιρροής. Και όταν θέτεται το ερώτημα γιατί μόνο οι πρώην κομμουνιστικές χώρες επλήγησαν από την κρίση αυτή του φυσικού αερίου. Αυτό είναι πολύ απλό να το απαντήσω. Γιατί λόγω ιστορικών λόγων εξαρτιόντουσαν σχεδόν αποκλειστικά από το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Απλώς έτσι έγιναν τα πράγματα ιστορικά. Η Ρωσία δεν είχε κάποιο σχέδιο να πιέσει την Σερβία ή τη Σλοβάκια, δεν ξέρω και εγώ ποια άλλη χώρα. <coughs> δεν έχουμε αρκετό χρόνο να συζητήσουμε τη διένεξη με την Ουκρανία για το φυσικό αέριο, αλλά νομίζω ότι δυστυχώς έχει παρερμηνευθεί αυτή η κρίση στην Δύση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ήταν μια τελείως διαφορετική κατάσταση από τις προηγούμενες περιστάσεις. Ήταν η πρώτη φορά που η Ουκρανία προσπάθησε να δείξει τη δύναμή της και να κρατήσει μια μονοπωλιακή θέση. Γι' αυτό η απόφαση Gazprom ή του Πούτιν να διακόψει την παροχή φυσικού αερίου ήταν ένα θανάσιμο σφάλμα, παρόλα αυτά ήταν αντίδραση στις ενέργειες της Ουκρανίας. Το ερώτημα τώρα του ποια σχέση θα ήταν πιο επωφελής, μια διμερής σχέση, μια σχέση της Ρωσίας με τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ως πολυμερής φορής. Η Ρωσία θα ήθελε να έχει περαιτέρω διμερή σχέση αυτή τη στιγμή βέβαια δεν γίνεται. Συγχρόνως είναι πάρα πολύ δύσκολο πολλές φορές να αντιμετωπίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν σύνολο. Γιατί ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμένες φορές έχει μια κοινή, ε, θέση και γνώμη, άλλες φορές όχι. Και υπάρχει και ε, μια διελκυνστίδα για την κατάκτηση αρμοδιοτήτων από την Κομισιόν έναντι των κρατών μελών και τούμπαλ. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να βρει κανείς αποτελεσματικές λύσεις για οποιοδήποτε εξωτερικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό περιλαμβάνει την Ρωσία. Σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ είναι ένας αρκετά ειδικό παίκτη. γιατί εμείς δεν κατανοούμε ποιος είναι ο μελλοντικός <clears throat> ρόλος του ΝΑΤΟ. Υπάρχει ένα ενοιολογικό πρόβλημα, γιατί το ΝΑΤΟ ακόμα δεν έχει μια στρατηγική αποστολή μετά από το τέλος του ψυχρού πολέμου. Για, για το λεγόμενο ανταγωνισμό σε επίπεδο γενεοδορίας. Ναι, και εγώ συμφωνώ στο ότι η Ρωσία δεν έχει καταφέρει καλά το να μπορέσει να προσελκύσει τις γειτονικές της χώρες. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ρωσική εξωτερική πολιτική και διπλωματία. Δυστυχώς δεν έχει γίνει ακόμα κάτι το οποίο να έχει αναγνωρίσει η, Σοβιετική, η, συγγνώμη, η ρωσική ηγεσία. Η Ρωσία για πολλούς λόγους αρχίζει τώρα να παρέχει κονδύλια στις γειτονικές χώρες οι οποίες έχουν θυγεί σοβαρά από την οικονομική κρίση. Ακόμα και για την Ουκρανία υπάρχουν σκέψεις να γίνει κάτι τέτοιο. Η άμεση αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι η Ρωσία καταχράται του οικονομικού του πλούτου προσπαθώντας να πιέσει να εξαγοράσει τις γειτονικές χώρες. Είναι τόσο λοιπόν ισχυρά και επίμονα τα στερεότυπα που πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς τι θα έπρεπε να κάνει η Ρωσία και τι δεν θα έπρεπε να κάνει. Η έννοια της σφαίρας επιρροής επίσης που ήρθε στη συζήτηση. Νομίζω ότι ήταν μία από τις χειρότερες δηλώσεις που έκανε στην διάρκεια της Προεδρίας του κ. Μετβέντεφ. Γιατί ήταν μία συγκινησιακή κατά κάποιο τρόπο αντίδραση στον πόλεμο της ε, Γεωργίας και αυτοί που θέλησαν να βάλουν την ιδέα των σφαιρών ε, ε, επιρροής μέσα στις πέντε βασικές αρχές της ρωσικής πολιτικής, μάλλον δεν σκέφτηκαν και πάρα πολύ τις συνέπειες. Βέβαια δεν έχει επαναληφθεί μια τέτοια δήλωση από τον πρόεδρο Μετβέντεφ ή τον πρωθυπουργό του κ. Πούτιν, προσπαθούν να αποφύγουν την μνήα των σφαιρών εφαρμογής. Αλλά αυτό ήταν μια ειδική στιγμή στον πόλεμο της Γεωργίας. Εγώ δεν θα ήθελα να εμπλακώ σε μια μακροσκελή συζήτηση για τη Γεωργία, αλλά το μόνο πράγμα το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης δεν έχει ολοκληρωθεί. Ήμασταν πολύ αισιόδοξοι πριν από 15-18 χρόνια όταν θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να γίνει με ειρηνικό και ανέμακτο τρόπο αυτή η κατάρρευση και ότι είχε ήδη ξεπεραστεί. Μιλάμε για ένα χώρο όπου υπάρχουν πολλά σοβαρά προβλήματα τα οποία θα ανακύψουν και πάλι επανειλημμένα. Δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό γιατί οι χώρες αυτές οι οποίες βρίσκονται στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και επί αιώνες επίσης στο ίδιο επίπεδο κρατικό δεν μπορούν να διαχωριστούν με τόσο μεγάλη ευκολία. Όλοι μας λοιπόν πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και ένας από τους λόγους από τα αίτια του πολέμου της Γεωργίας ήταν ακριβώς η επιθετική πολιτική που ακολουθήθηκε από την προηγούμενη Αμερικανική κυβέρνηση. Κάτι ακόμα. Η Ρωσία έχει διαδραματίσει ένα διαφορετικό ρόλο στον ε, Νότιο Κάυκασο την εποχή, από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Αλλά και οι τέσσερις κύριοι πόλεμοι στην Γεωργία έχουν ξεκινήσει από τη γεωργιανή πλευρά. Μπορούμε να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες, αλλά και στις τέσσερις περιπτώσεις η γεωργία ξεκίνησε τις εχθροπραξίες. Τέλος, τα θέματα ενέργειας. Οι χώρες οι οποίες παράγουν ενεργειακούς πόρους δεν έχουν μέλλον, όπως είπε κάποιος προηγουμένως. Θα αλλάξει η κατάσταση στον ενεργειακό τομέα. Αληθεύει αυτό και η Ρωσία φυσικά δεν μπορεί να αποφύγει τη μεταρρύθμιση των οικονομικών της δομών εάν θέλει να παραμείνει ένα σημαντικός παίκτη σε διεθνές επίπεδο. Αλλά συγχρόνως θέλω να σας υπενθυμίσω ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αλλάξει την αντιμετώπιση της σε πολιτικό επίπεδο αν πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να παραμείνει σε ηγητικό επίπεδο στον 21ο αιώνα. Γιατί η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει να παριστάνει ότι μπορεί να ζήσει μέσα σε μια γυάλινη σφαίρα, σε ένα απομονωμένο απομονωμένη από το διεθνές πλαίσιο και τις δυνάμεις που δρούν στο διεθνές θερέωμα. Βλέπουμε να υπάρχει στο διεθνή χώρο όλο και αυξανόμενος ανταγωνισμός ακόμα και σε επίπεδο στρατιωτικών δυνάμεων που έχουν επανέλθει στο διεθνή χώρο. Είναι πολύ ωραία η εικόνα αυτή που λέει ότι η Ευρώπη έχει μονάχα ήπια δύναμη που είναι πολύ καλύτερη από την σκληρή δύναμη, τη στρατιωτική. Αλλά οι ελπίδες που είχαμε στη δεκαετία του 1990 ότι θα άλλαζε η μορφή του διεθνού συστήματος δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Και στο μέλλον, για να μπορέσει να διαδραματίσει κάποιο ρόλο, ο κάθε παίκτη σε διεθνείς, σε διεθνείς συνθήκες θα χρειαστεί και ήπια αλλά και σκληρή δύναμη, κάτι το οποίο αποτελεί ένα πρόβλημα με την ε, ε, Ευρώπη. Για τον κύριο Γιακυμένκο, εδώ διαφωνώ με τον κύριο Κόζατσεφ. Ο κύριος Γιακυμένκο, ο οποίος ήταν ο πρώην ηγέτης της εθνικής κίνησης στη Ρωσία, είναι το πιο άσχημο πρόσωπο της ε, μετασοβιετικής εξέλιξης στη Ρωσία. Δεν νομίζω λοιπόν ότι έχει κάποια σχέση με την Ευρώπη, δεν έχει κάτι να προσφέρει στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Uh, ευχαριστώ πολύ κύριε Λουκιάνοφ, ευχαριστώ όλα τα μέλη του πάνελ. Το δεύτερο πάνελ θα καταλήξει στα συμπεράσματά του. Να πω μερικά λόγια, αναφερθήκαμε στις σχέσεις. Ούτε στατική ούτε απλή είναι η σχέση με τη Ρωσία, αυτό το συμπέρασμα και θα πρέπει να είναι σοβαρή όπως είπε κάποιος και ευφυής όπως είπε κάποιος άλλος. Το πρώτο πάνελ έκανε τη διάγνωση. Το δεύτερο πάνελ αφορά το μέλλον. Καλό τα μέλη του δεύτερου πάνελ να έρθουν εδώ στο βήμα. Спасибо.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 Κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε, έχουμε μείνει πίσω, αλλά αυτό σημαίνει ότι το θέμα είναι και ενδιαφέρον και χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Και, όπω και όπως είπε ο Κωνσταντίνη Κωνστατσόφ, χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο και περισσότερες ευκαιρίες ε, για συζήτηση. Περνάμε λοιπόν στο δεύτερο πάνελ. Το μέλλον των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ενώσεως Ρωσίας και είναι κάτι παραπάνω από ενεργειακό ζήτημα. Ο τα μέλη του πάνελ είναι ο κ. Άντος του Ινστιτούτου Πέτερσον για τη Διεθνή Οικονομία που εξοικειδεύεται στην οικονομική πολιτική Ρωσία, Ουκρανία και Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και ήταν οικονομικός σύμβουλος για τι κυβερνήσει Ρωσία, Ουκρανίας και Κυριστάν ήταν διευθυντή του Ινστιτούτου Στοχόλμη για μεταβατική οικονομία και καθηγητή στην σχολή, οικονομική σχολή τη Στοχόλμη. και ήταν και διπλωμάτη στη Μόσχα, στη Γενέβη και στο Κουβέιτ και συνέγραψε εννέα βιβλία, έγραψε αυτόν το τελευταίο πώ η Ουκρανία έγινε οικονομία τη αγορά και δημοκρατία και δεν έχει ερωτηματικό τίτλο. εξεβονίμων Άντριο Βίλσον στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ξένων ε, σχέσεων, ε, Εξωτερικών Σχέσεων από το University College του Λονδίνου και το Royal Institute of International Affairs και ο Ίγκο Πουπέσκου αριστερά του από τη Μολδαβία, αυτή είναι η υπηκότητά του, είναι, ζει στο Λονδίνο, διδάσκει την ε, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πολιτική γειτονίας, με τις ανατολικές χώρες και, και διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο της ε, Βουδαπέστης. Τα μέλη του ΠΑΝΕ, λοιπόν ζητήσαμε τις υπηρεσίες μας να μας πούν κατά πόσο θα ξεπεράσουμε τα όρια μας, ναι. Θα δουλέψουμε μέχρι μία, λέει ο πρόεδρος, και όχι 12 και 30, λέει διατείνεται ο πρόεδρος. Ο κ. Άστον έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή για μένα που είμαι εδώ ξανά και όποτε ο κύριος Σάριου Βόλσκι με καλεί στην Ευρώπη πάντα μπαίνω στο αεροπλάνο και έρχομαι στις Βρυξέλλες γιατί είναι μεγάλη τιμή για μένα γιατί ξέρω ότι πάντα οι συζητήσεις εδώ είναι πολύ καλές και ενδιαφέρουσες όπως είδαμε σήμερα το πρωί. Μου ζήτησαν σήμερα να μιλήσω για το θέμα το εξή. Ρωσική οικονομία, κάτι παραπάνω από ενέργεια και διάλεξα τρία θέματα που θα συζητήσω μαζί σας. Το πρόβλημα της ενέργειας, η παγκόσμια οικονομική κρίση και η κρίση για το φυσικό αέριο. Το μεγάλο θέμα. Πρώτα απ' όλα πόσο σημαντική είναι η ενέργεια για τη ρωσική οικονομία. 65% των εξαγωγών της Ρωσίας πέρσι 50% περίπου του κρατικού εισοδήματος αλλά μόνο 20% του ΑΕΠ. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι 45% του ΑΕΠ της Ρωσίας προέρχεται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Ρωσία έχει 8,4 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις καταχωρημένες. Οπότε η πυκνότητα των επιχειρήσεων είναι περίπου ίση με αυτή της Δυτικής Ευρώπης αλλά αυτή η σημασία αυτών μειώθηκε τελευταία χρόνια. Η υψηλή τιμή του πετρελαίου μετά το 2004 επέτρεψε στον Πούτιν να εφαρμόζει κάποια μέτρα και άλλαξε η κατάσταση. Θα μπορούσε να έχει αυτή η εικόνα είναι από την προσωπική του ιστοσελίδα. Αν έτσι θέλετε, θέλει να παρουσιάζεται. Mm. Εδώ, ένστολος. Λοιπόν, ε, έχουμε προβλήματα διαφθοράς, ε, παρεμβατισμού του κράτους κλπ. Η Gazprom αποφάσισε να κάνει περικοπές στην παραγωγή φυσικού αερίου κατά 8%. Και έτσι δρά ένα μονοπόλιο. Και η διαφθορά είναι εκτός ελέγχου. Ε, είναι σε θέση 147 η Ρωσία από τις 180 χώρες όσον αφορά την διαφάνεια. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν χώρες που είναι πλουσιότερες από τη Ρωσία. Μόνο ε, η σημερινή Γουινέα είναι πλέον διαφθαρμένη από τη Ρωσία. Δεν είναι καλή αυτή η εικόνα και η θέση για τη Ρωσία. Και έχει συνέπειες αυτό μετά το 2000 δεν έχει κάνει συντήρηση του δικού δικτύου της και να το αναπτύξει. Είναι πολύ διεφθαρμένη η Ρωσία για να εκτελέσει έργα υποδομών. Και έχει μείνει εκτός η Ρωσία και για άλλο λόγο. Είναι πολύ πλούσια και θα έπρεπε να είναι ανοιχτή. Δεν έπρεπε να είναι τόσο αυταρχικό το κράτος στη Ρωσία και νομίζω ότι το φαινόμενο αυτό ε, της μεγάλης αυταρχικότητας είναι προσωρινό. Μόνο μία νομιμότητα, κάτι, μόνο κάτι σωστό είχε το καθεστώς Πούτιν, μεγάλο ρυθμό οικονομικού ανάπτυξης. Μόνο χαμηλή τιμή του πετρελαίου και της ενέργειας μπορεί να θέσει κίνδυνο το καθεστώς Πούτιν. Και είναι πολύ ευάλωτη στην οικονομική κρίση η Ρωσία σήμερα. 85% των εξαγωγών είναι βασικά προϊόντα της Ρωσίας, αλλά εξαρτάται από τις τιμές. Μπορεί να μειωθούν 40% φέτο εξαγωγές, χάλιβας, οικοδομές, χημική βιομηχανία ε, ή θα μείνει σταθερή κατάσταση ή κατά μισό, μισή, μισή ποσοστία μονά θα μειωθεί, άρα και το ΕΠ θα μειωθεί πιθανότατα. Το τραπεζικό σύστημα είναι, ε, αντιμετωπίζει προβλήματα, διότι κυριαρχούν οι κρατικές τράπεζες το κράτος βγάζει τα χρήματα στο εξωτερικό μέσω ε, από τα αποθέματα συναλλάγματος. Και τελικά όλα αυτά δεν τα θέλουμε σε μια οικονομική κρίση διεθνή. Έχουν, υπάρχουν σοβαρές συνέπειες λόγω όλων αυτών που γίνονται. Τα αποθέματα μειώθηκαν κατά 210 δις δολάρια το συναλλαγματικό απόθεμα η πολιτική αντιμετωπίσεως της κρίσης. Ξεκίνησε τέτοια πολιτική η Ρωσία τον Οκτώβριο, τον περασμένο. Δεν πέτυχε όμως πολλά. Μόλις πριν από 15 μέρες ο Πρωθυπουργό ο Βλαντιμίρ Πούτιν που είναι και ο βασικός οικονομολόγος της Ρωσίας παραδέχτηκε ότι αντιμετωπίζει οικονομική κρίση η χώρα. Το αρνεί το επί Μακρόν ο Πούτιν και κατηγόρησε τη ΣΥΠΑ για την κρίση κατηγορούσε μάλλον. Δεύτερον, ο πρόβλημα μπορεί να χρησιμοποιήσει την κρίση για την εθνικοποίηση αρκετών επιχειρήσεων. Και τελικά θα κρατικοποιηθούν δύο μεγάλες επιχειρήσεις χωρίς βάσιμους λόγους. Και μετά προσπαθεί, ε, όλοι έχουν καταλάβει ότι η ισοτιμία τελικά θα μειωθεί και γίνεται κερδοσκοπία εναντίον του ρουβλιού και όταν τυπώνει ε, και άλλα χρήματα η κεντρική τράπεζα τα αλλάζει ο κόσμος για περισσότερα δολάρια. Οπότε 80% ε, μειώθηκε, ε, μειώθηκαν οι συναλλαγές στο χρηματιστήριο. Άρα, ποιες είναι οι συνέπειες. Η οικονομική κρίση ε, έχει εξίσου σημαντικές συνέπειες στη Ρωσία όπως και αλλού στον υπόλοιπο κόσμο. Το ΑΕΠ μειώνεται και οι επενδύσεις μειώνονται. Σημαντικά βιομηχανική παραγωγή τώρα καταραίει, 10% έχει μειωθεί το Δεκέμβριο και το πραγματικό εισόδημα που αυξανόταν σημαντικά με ρυθμούς 13% το χρόνο για πολλά χρόνια τώρα μειώθηκε κατά 12% το Δεκέμβριο. Λοιπόν, ποια είναι τα συμπεράσματα. Ο Πούτιν ήταν τυχερός, αλλά έκανε λίγα πράγματα για τη Ρωσία. Το αυταρχικό καθεστώς του είναι εύθραυστο και αυτό σημαίνει ότι το status quo δεν αποτελεί επιλογή σήμερα. Είναι σαν σταυροδρόμι η Ρωσία. Δύο επιλογές έχει. Ή μεγαλύτερο αυταρχισμό με κρατικό καπιταλισμό και προστατευτισμό και δεν χρειάζεται συνεργασία με Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την περίπτωση ή θα δούμε μια πολιτική και οικονομική ε, φιλελευθεροποίηση που είναι διαφορετική, αντίθετη κατεύθυνση. Τώρα πάμε στον πόλεμο του φυσικού αερίου και θα αναφερθώ ακροθυγώς στις συνέπειες αυτού. Ε, καλή συμφωνία, δεν υπάρχει μεσάζων, είναι μακροπρόθεσμη συμφωνία, κανονικές τιμές και δασμοί καθορίζονται μέσω τύπου. Είναι βασικά μια νίκη για την Ουκρανία αυτή αυτή η συμφωνία συνήφθη 31 Δεκεμβρίου. Δεν υπήρχε λόγος για το πόλεμο του φυσικού αερίου, κανένας λόγος. Υπήρχε συμφωνία. Δείτε την εικόνα από τις διαπραγματεύσεις 17 με 18 Ιανουαρίου τα λέει όλα η φωτογραφία από την σελίδα της Τζούλια Τιμοσέγκο. Εδώ συναντώνται και βλέπετε ότι είναι συνάντηση επιχειρηματική, συνομιλιών οικονομικών και σπάνια βλέπετε τον Πούτιν τόσο χλωμό και αυστηρό, κυρίως μετά την λήξη των διαπραγματεύσεων. Βλέπετε ότι η Τζούλια Τιμοσέγκο έχει ψηλά το κεφάλι και ο Πούτιν φαίνεται πολύ δυστυχής. Λοιπόν, 19 Ιανουαρίου τα πρόσωπα των διαπραγματευτών. Πολύ σπάνια βλέπει κανείς τον Πούτιν τόσο τρομαγμένο και δυσαρεστημένο. Η καλύτερη φωτογραφία. Κοιτάξτε το πρόσωπο του Πούτιν. Ποιες είναι οι συνέπειες για την Ουκρανία. Η Ουκρανία τώρα έχει προβλέψιμους όρους για τις παραδόσεις φυσικού αερίου και την τιμολόγηση. Ήταν τεράστια πηγή ε, διαφθοράς και πολιτικής χρηματοδότησης. Άρα μεγαλύτερη εξαρτησία από τη Ρωσία και την Ουκρανία. Για την Κάσπρομ. οι συνέπειες είναι αρκετά καταστροφικές. Πώς μπορεί ποτέ ε, να αποδείξει ότι είναι αξιόπιστος προμηθευτής η Κάσπρομ. δεν μπορεί πια και οι μετοχές της έπεσαν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Οι συνέπειες για τη Ρωσία. Ε, μειώθηκε η φήμη της, ε, επιβλαβής η φήμη της, ε, βλάφτηκε η φήμη έγινε αναξιόπιστη, έχασε την επιρροή της επί και τελικά, τελικά ενώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι αυτής. Ποιες είναι οι συνέπειες για την Ευρωπαϊκή Ένωση προφανή τα συμπεράσματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια ενεργειακή πολιτική, χρειάζεται αποσύνδεση των διαφόρων κλάδων της παραγωγής, της μεταφοράς και της πωλήσει, χρειάζεται μεγαλύτερο αποθεματικό. Η Ουκρανία χρησιμοποιεί πολύ καλά τα αποθέματα, δεν υπέφερε γι' αυτό. Χρειάζεται περισσότερο υγραέριο, μεγαλύτερη ποικιλομορφία όσον την ενέργεια. Βλέπουμε αρκετέ χώρε όπως η δική μου γενέτειρα, η Σουηδία και η Πολωνία, που εξετάζουν θετικότερα την πυρηνική ενέργεια και βεβαίω χρειάζεται μεγαλύτερη αλληλεγγύη όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια πολιτική για τη Ρωσία, χρειάζεται ένα ενωμένο μέτωπο, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι κάθε χώρα ξεχωριστά Ευρωπαϊκή Ένωση να διαπραγματεύεται. Ήταν συγκινητικό που ακούσαμε ότι ο Βλαδιμίρ Πούτιν διαμαρτυρήθηκε ότι η Ουκρανία δεν συμμορφώθηκε με την ενεργειακή χάρτα ενώ η Ρωσία δεν την ε, κύρωσε. Υπέροχη δυνατότητα να αναζωογονηθεί η χάρτα η ενεργειακή και η Ρωσία να ε, συμμετάσχει περισσότερο και ενταχθεί σε αυτό το πλαίσιο. Υπήρχαν και άλλες συνέπειες για την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι χρειάζεται να κατασκευάσει τον Αμπούκο όπως είπε και το προηγούμενο πάνελ Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ζητήσει ή να κάνει μεταρρυθμίσεις ενεργειακές η Ουκρανία, ούτως ώστε να απαλλαγεί από τις διεφθαρμένες πρακτικές. Και αυτό θα πρέπει να απαλλαγει απο τις διαθαρμενες πρακτικες και αυτο θα πρεπει να συμπληρευτει συμφωνία σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και τελευταίο σημείο που θέλω να θίξω είναι ότι είναι σημαντικό να υποστηριχθεί η σταθεροποίηση της Ουκρανίας μέσω πιστώσεων διεξάγεται μια συζήτηση τώρα μεταξύ Πούτιν και Τιμοσέγκο να δώσει η Ρωσία 5 δισεκατομμύρια δολάρια για πίστοση σταθεροποίησης προς την Ουκρανία. Βασικά αυτό δεν είναι προβληματικό, αλλά δεν θα πρέπει να προέρχονται χρήματα μόνο από τη Ρωσία και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δώσει ανάλογες πιστώσεις. Χρειάζεται συγχρηματοδότηση, ήθιστε. Συμφωνίες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου η Ευρωπαϊκή Ένωση το έκανε αυτό για την Ουγγαρία και για τη Λετωνία. Νομίζω ότι θα ήταν καλό αυτή η πρακτική να επεκταθεί και στην περίπτωση της Ουκρανίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you, Mr. Uh, ευχαριστώ. Ε, παρουσιάσατε το θέμα σας με τη γνωστή σας ε, ευφυΐα και διορατικότητα. Θα περάσουμε στην επόμενη παρουσίαση τώρα του κύριου Ουίλσον. Είναι δύο συν, συντάκτες αν θέλετε. Έχετε το λόγο εσείς κύριε Ουίλσον. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας. Το έγγραφό μου θεωρεί ότι υπάρχουν δύο σημαντικά θέματα. Αλληλεγγύη και κράτος δικαίου. Στο έγγραφο εξετάζουμε πώς μπορούν να ε, εφαρμοστούν σε τέσσερις διαφορετικούς τομείς. Πρώτο, ποια πρέπει να είναι η προσέγγιση μας προς τη Ρωσία. Ο πόλεμος στην Γεωργία οδήγησε σε, κάποια, σε κάποιο απομονωτισμό αλλά χωρίς ε, να υπάρχει συνένεση από πλευράς ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης για ε, αυτή την απομόνωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να στοχεύσει να συνεχίσει να εξάγει ευρωπαϊκές αξίες όχι θεωρώντας ότι αυτές είναι οι κοινέ. Η πρόθεση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, της ελεύθερης οικονομίας της αγοράς κτλ. θα χρειαστεί κάποια προσπάθεια και θα χρειαστεί και πόρους. Η προσέγγιση κράτους δικαίου σημαίνει να ασκηθεί η πίεση για να υπάρξουν πραγματικές αλλαγές στη Ρωσία. Όπως είπε ο πρόεδρος Μετιέντες στην αρχή της προεδρίας του. Και οι απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την ε, Ρωσία θα πρέπει να είναι πιο συνεπείς. Έμφαση στο κράτος δικαίου σημαίνει και σύγκληση των ευρωπαϊκών συμφερόντων και των χωρών μελών. Και τέλος θα προσφέρει και πιο αποτελεσματικό τρόπο ε, για να μιλεί η Ευρώπη στην ε, Ρωσία, ε, ζητώντας να, δεσμευ... να τηρήσει τις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις της προκύπτουν από τη συμμετοχή της στο Συμβούλιο της Ευρώπης κλπ. Δεύτερο τώρα, αλληλεγγύη και κράτος δικαίου θα πρέπει να αποτελέσουν την βάση για εσωτερική αλληλεγγύη που θα αποτελέσει και το κριτή για οποιαδήποτε αποτελεσματική εξωτερική ρωσική πολιτική προς τη Ρωσία δηλαδή. Όπως ε, φάνηκε και στην κρίση της Γεωργίας και του φυσικού αερίου, οι διμερείς ε, συζητήσεις μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών και της ε, Ρωσίας έχουν μπλοκάρει τον ευρωπαϊκο-ρωσικό διάλογο. Από την άλλη μεριά, οι διμερείς συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής, ευρωπαϊκών χωρών και Ρωσίας υπονομεύουν την αλληλεγγύη και έχει γίνει και κατάχρηση των βέτο. Θεωρούμε λοιπόν ότι το πρώτο βήμα για την αποτελεσματική εφαρμογή μιας εσωτερικής αλληλεγγύης στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι και η αμοιβαία, βασισμένη στην αμοιβαία ευθύνη των χωρών μελών απέναντι των μεν δε. Και μια εταιρική σχέση που να οδηγήσει και σε σημαντικέ πρωτοβουλίε στην εξωτερική πολιτική. Εξηγούμε και ορισμένου μηχανισμού για να λειτουργήσει η αλληλεγγύη στην πράξη. Ε, Όπω με ευρωπαϊκέ αποστολέ αξιολόγηση στι ε, χώρε όπου συμβιώνονται διαμάχε κλπ. Τρίτο, οι ίδιε αρχέ πρέπει να διέπουν και τι ε, προσπάθειε τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην ε, κοινή πολιτική γειτονία. Πρώτα, η πολιτική γειτονία είναι ανταγωνιστική. Δεν έχει αναγνωρίσει εύκολα η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ότι υπάρχει ε, μια ανταγωνιστική, ανταγωνιστική σχέση με τη Ρωσία. Δεν είναι όμω ανταγωνισμό σφαιρών επιρροή η ε, προσπάθεια πολιτικού ελέγχου τη περιοχή. Είναι ανταγωνισμό που ανταποκρίνεται περισσότερο στι ατομικέ ανάγκε των μελών και ανταγωνισμό μεταξύ πολιτικών και οικονομικών μοντέλων που προσφέρονται στου γείτονε. Ρωσία μπορεί να χρησιμοποιήσει την κρίση της Ρωσίας προσωρινά για να κάνει πιο σαφή την πολιτική της αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να προσπαθήσει να αποκτήσει μια δική της σφαίρα επιρροής, αλλά να προσφέρει τη δυνατότητα στις χώρες της πολιτικής γειτονίας να αναπτύσσουν τις δικές τους επιλογές. Δεύτερο, πρόκειται για κυρίαρχη γειτονία. Είναι αδύναμες χώρες και για αυτές το να δημιουργήσουν ισχυρά κράτη είναι προτεραιότητα. Χωρίς απαραίτητα να είναι η προτεραιότητά τους να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για να το κάνουν αυτό, κάνουν προσπάθεια εξισορρόπησης της κατάστασης μεταξύ ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Σε μια προσπάθεια να υιοθετήσουν και ένα μέρος του κοινωτικού και εκτιμένου. Και τρίτο, η γειτονία η οποία ήδη είναι αδύναμη, έχει ε, τρωθεί και πολύ από την οικονομική κρίση. Προσπαθώντας να φτιάξουν κυρίαρχα κάτι, οι ε, χώρες αυτές της πολιτικής γειτονίας έχουν ε, αγνοήσει άλλα σημαντικά καθήκοντα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει βοηθήσει επαρκώς για να ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτές. Στα 90 το μοντέλο ήταν περισσότερο προσφορά από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξαγωγή του κοινοτικού κεκτημένου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνοντας ιδιαίτερη, ε, κάνοντας ιδιαίτερη προσπάθεια για την ενίσχυση των θεσμών της και για την αύξηση τη απορροφητικότητά τη. και μια πολιτική γειτονία η οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τι ιδιαίτερε αδυναμίε τη κάθε χώρα, η οποία εντάσσεται σε αυτήν. Στο έγγραφό μα. αναφερόμαστε σε έξι ξεχωριστές ε, προσεγγίσεις στρατηγικής για κάθε μια από τις έξι χώρες. Και τέλος, εμείς λέμε πέραν της πολιτικής ενέργειας, αυτό είναι ο τίτλος του εγγράφου μας. Όμως οι ίδιες αρχές αλληλεγγύης και κράτους δικαίου εφαρμόζονται και στον τομέα της ενέργειας. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να αναπτύξει μια πιο συνεκτική πολιτική απέναντι στη Ρωσία, πρέπει ε, να ε, προσέξει και ιδιαίτερα τον τομέα τη ενέργεια και του αερίου. Και πριν από την κρίση του Ιανουαρίου ήταν σαφέ τι πρέπει να γίνει. Τώρα όμω υπάρχει περισσότερη πολιτική βούληση για ανάληψη δράση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει σημαντική πρόοδο για να εξασφαλίσει μια ενιαία και λειτουργική αγορά του φυσικού αερίου για την εξασφάλιση της ασφάλειας προμηθειών και να δείξει αλληλεγγύη στη, στην επόμιση των βαρών. Είναι σε μια πραγματική διεθνοποίηση του συστήματος αγωγών διαμετακόμισης του φυσικού αερίου. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορεί να γίνει αυτό. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιλέξει να παρακάμψει την ε, Ουκρανία, θα χάσει αλλού. Οι πρώην χώρε διαμετακόμισης είναι ήδη αδύναμε και οι οποίοι θα παρακαμφθούν δηλαδή και θα γίνουν ακόμη πιο αδύναμε. Δεύτερο, η Ουκρανία <coughs> δεν θα μπει σε ένα διεθνοποιημένο σύστημα αγωγών εφόσον ε, στην ουσία διαχειρίζεται τα θέματα της η Gazprom. Η Ουκρανία είχε την αίσθηση για την κρίση του Ιανουαρίου ότι βρισκόταν ε, μεταξύ Σκύρας και Χαρίβδος όπου και τα δύο πλευρές είναι Gazprom. Θα πρέπει να υπάρξει και μια ε, συνθήκη για την ασφάλεια της ε, παροχής φυσικού αερίου με προβλέψεις για την ε, επίλυση διαφωνιών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Βίλσον. Περνάμε στη, συζήτηση τώρα. Ο κύριος Γκίρτιχ θα έχει το λόγο. Θέλω καταρχήν να σχολιάσω αυτά που είπε ο κύριος Λιουκάνοφ. Νομίζω ότι εξακολουθεί να έχει εγκυρότητα θα από αυτό το οποίο ήθελα να πω. Ανέφερε ότι η Ρωσία και η Ευρώπη είναι πολιτιστικά πολύ κοντά. Εγώ το διαμφισβητώ αυτό. Υπάρχει πολιτισμική διαφορά μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας που δεν μπορεί να αγνοηθεί αν πρόκειται να είναι καρποφόρες η σχέση μας. Εμείς έχουμε διαφορετική κατανόηση της δημοκρατίας. Στη Ρωσία όλα βασίζονται στο ότι ο λαός ψηφίζει υπέρ του τσάρου. Αλλά το θέμα είναι ποιος είναι ο τσάρος. Ξέρουμε τις διαφορές μεταξύ Ευρώπης και Σαουδικής Αραβίας. Καμιά από τις δύο πλευρές δεν προσπαθεί να αλλάξει την άλλη. Είναι καλές οι σχέσεις γιατί αναγνωρίζονται και γίνονται αποδεκτές οι διαφορέ, Το ίδιο πρέπει να γίνει και σε σχέση με τη Ρωσία. Πρέπει να αποδεχτούμε το γεγονός ότι είμαστε διαφορετικοί σε πολιτισμικό επίπεδο και να σταματήσουμε να προσπαθούμε να αλλάξουμε ο μεν, τον δε και τούμπαλιν. Να σταματήσουμε να θέλουμε να κάνουμε τις πολιτικές και οικονομικές σχέσεις εξαρτημένες από μια αλλαγή ταυτότητα. Όλοι οι πολιτισμοί θέλουν να επεκταθούν. Είναι φυσιολογικό αυτό, λέει. και πολιτικέ και σχέσεις θα πρέπει να παραμείνουν χωριστές από τις ελπίδες επέκτασης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τάνοκ, αντιπρόεδρος της αντιπροσωπείας με την Ουκρανία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να χαιρετήσω θερμά το πάνελ, ιδιαίτερα τον Άντερς Άσλαντ. Κύριε Πρόεδρε, σε εσάς μιλάω. Γεια σε εσένα λέω γράψαμε ένα άρθρο μαζί για το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας, το οποίο δημοσιεύτηκε. Δεν ξέρω αν ο Άντερς θα έχει το θάρρος να σχολιάσει το... την είδηση που πήρα σε μια συνάντηση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας ο πρόεδρος Ιουσένκο στην Ουκρανία έκανε μια μεγάλη επίθεση εναντίον ενός πρωθυπουργού που δεν μπορεί τώρα να απολύσει χωρίς εκλογές αλλά περιέγραψε τη συμφωνία για το φυσικό αέριο που αναφέρατε ως ένα σύμφωνο Ρίμπεντροπ Μόλοτοφ, ως μια παραχώρηση, ως ένα ξεπούλημα προς την, για την Ουκρανία. Είναι, δεν ξέρω αν αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να δει κανεί ω κάτι διαφορετικό από μια επίθεση προς την Πρωθυπουργό του, γιατί αυτό δεν είναι ανταποκρίνεται και προς την αλήθεια. Φαίνεται ότι ήταν μια πολύ καλή συμφωνία. Μια συμφωνία που ήταν μεγάλο βάρος για την ε, Ουκρανία, η οποία έχει ξεπεραστεί πλέον. Επίσης, <clears throat> για το θέμα αυτό, που, για ένα θέμα που είναι σχετικό. Εγώ ενοχλούμε συνέχεια για την απόκληση μεταξύ αυτών των δύο ηγετικών προσωπικότητων στην Ουκρανία. Είναι καιρός ο πρόεδρος να μπορέσει να εξασφαλίσει μια ενότητα στην εξωτερική εικόνα της Ουκρανίας με το να ξεπεραστεί το θέμα αυτό με την Πρωθυπουργό του. Αναρωτιέμαι αν η Τσεχική Προεδρία, και το έθεσα Χθε θα μπορούσε να καλέσει και την κυρία Τιμοσέγκο και τον πρόεδρο Γιουσέγκο στη μεγάλη συνδιάσκεψη που θα γίνει το Μάρτιο για τα θέματα της εταιρική σχέσης με την Ανατολική γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως θα πρέπει λοιπόν να αφήσουν κατά μέρος τις εσωτερικές τους διαφορές οι ηγέτες της Ουκρανίας και να δουν το ρόλο της Ουκρανίας στο διεθνή στίβο. Ευχαριστώ κύριε Τάνοκ. Ο Κρίστοφερ Μπίστλεϊ, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για τη Βαλτική Στρατηγική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζήτω και συγγνώμη που δεν μπόρεσα να με πάρουν στο σύνολο της ακρόασης. Απλώς θα ήθελα να σταθώ λιγάκι σε αυτό το οποίο ανέφεραν προηγουμένως οι συνάδελφοι για το αν έχει αλλάξει ή αν αλλάζει κάτι στις σχέσεις Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μια διαφορετική αμερικανική κυβέρνηση, ο Τζο Μπάιντεν το ανέφερε και αυτό προς τους Ρώσους συναδέλφους. Ο κύριος Ιβανοφ, θυμάμαι, είχε δώσει δύο συνεντεύξεις στο Russia Today και στο CNN για το ίδιο θέμα, για την ίδια συνάντηση, δίνοντας διαφορετικές <clears throat> πληροφορίες στο CNN από στους Ρώσους, στο Russia Today. Στο CNN είπε μια χαρά πήγαν όλα, έχουμε φτιάξει πολύ καλές σχέσεις. Στο Russia Today είπε είδα να υπάρχει μια βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας στο παρελθόν, αλλά έρχονται και φεύγουν αυτές οι αλλαγές. Δεν πιστεύω θα υπάρξει ουσιαστική αλλαγή. Αναφέρθηκε ο Τσάρος από τον κύριο Ζήρτη. Αλλά ο Πρωθυπουργό είναι αυτός ο οποίος ασχολείται με τα θέματα εξωτερικών υποθέσεων και ασφάλειας. Δεν βλέπω κάποια ένδειξη για το ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα αλλάξει τις απόψει του σε σχέση με τις εξωτερικές σχέσεις της Ρωσίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή με οποιαδήποτε άλλη κυριαρχή χώρα. Γιατί νομίζω ότι η με οποιαδηποτε αλλη κυριαρχη χωρα γιατι νομιζω οτι η νοτροπια που επικρατεί είναι ότι ναι, δεν έχουμε τη Σοβιετική Ένωση πλέον, αλλά θα ασκήσουμε την επιρροή μας χρησιμοποιώντας τους ενεργειακούς μας πόρους για να μπορούμε να έχουμε έλεγχο, επιρροή και ισχύ στην πρώην Σοβιετική Ένωση ή αν θέλετε στην πρώην Ρωσική Αυτοκρατορία. Είναι λοιπόν ζωφερή η εικόνα και σε ό,τι αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαιρέσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δυτικοευρωπαίοι, όπως μας θυμίζουν οι ανατολικοευρωπαίοι συναδελφοί μας, έχουν την αφελή άποψη ότι αρκεί να πάμε στη Ρωσία να υπογράψουμε μερικέ συνθήκε και θα είναι όλα με λιγάλα. Ενώ οι Ανατολικοευρωπαίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να είναι βαθιά καχύποπτοι σε σχέση με τι προθέσεις της Ρωσία. Το ερώτημα μου λοιπόν είναι, έχει αλλάξει κάτι στη Ρωσία. Από την τελευταία φορά που εξετάσαμε αυτό το θέμα την εποχή του πολέμου της Γεωργίας ή απλώς επιδεινώνται οι σχέσεις μας έκτοτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπίσλε. Ο κύριος Ονισκίεβιτς. Ευχαριστώ. Έχω κάποια ερωτήσει για τον κύριο Όστλουντ. Πρώτα απ' όλα, ποιες είναι οι πηγές των ρωσικών οικονομικών προβλημάτων, ποια είναι τα αίτια, συνδέονται μόνο με τη γενική χρηματοπιστική κρίση διότι υπάρχουν ενδείξεις ότι το πρόβλημα αυτό άρχισε πριν ξεσπάσει η χρηματοπιστωτική κρίση. Δεύτερον, σε ποιο βαθμό μπορούμε να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι η Gazprom μπορεί να ανταποκριθεί στις συμβατικές της υποχρεώσεις όσον αφορά την παροχή πετρελαίου και φυσικού αερίου χωρίς την εισρωή ξένου κεφαλαίου στο πάνω κομμάτι της αλυσίδας ή στην παραγωγή. Διότι θεωρούμε πολύ ότι η Gazprom βγήκε για ψώνια. Ξόδεψε πολλά χρήματα για να αγοράσει αγωγούς και να αγοράσει συστήματα διανομής και δεν επένδυσε αρκετά στην παραγωγή. Και νομίζω ότι της λείπουν περίπου 60 με 80 κυβικά... εκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο για να αποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Σήμερα. Τι θα γίνει στο μέλλον. Και η προσχώρηση στον ΠΟΕ και η αύξηση των τιμών ενέργειας στο εσωτερικό της χώρας τι συνέπειες έχουν για την οικονομία της Ρωσίας. Ευχαριστώ. Ο κ. Πρίμπετης των Σοσιαλιστών έχει το λόγο κύριε Πρόεδρε. Euh, ναι, ναι, ναι, Τώρα όσον αφορά την ανεξαρτησία, αφού χαιρετήσω βέβαια τα όσα είπαν οι προϊολαλήσαντες, ο καλύτερος τρόπος να είναι κανείς ανεξάρτητος είναι να μην εξαρτάται πλέον. Σοφιστία βέβαια αυτή. Η κρίση του πετρελαίου βασίστηκε στην ανάγκη να εξασφαλίζεται η ασφάλεια προμήθειας μάλλον. Μας οδήγησε μετά από την κρίση του πετρελαίου και πολλές χώρες του, της πρώην Σοβιετικής Ένωσης πιάστηκαν ήδη από το λαιμό και πνίγονται από την κρίση λόγω ελλείψεως ρευστότητα και δυνατότητας ε, παροχής ενέργειας. Για τους Γάλλους, όπως και για άλλους, κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης του 1974, η πυρηνική ενέργεια αναπτύχθηκε για να υπάρχει πραγματική ανεξαρτησία. Και διαρωτώ μετά από την κρίση του φυσικού αερίου και λόγω της συμπεριφοράς της Ρωσίας, διερωτώ με, η Ρωσία μήπως ξεκίνησε όχι οκτωβριανή επανάσταση ενεργειακή, αλλά απλή επανάσταση. Διότι υπεύθυνοι οι Ευρωπαίοι διερωτώνται να στραφούν προς καλύτερη ανεξαρτησία προσπαθώντας να αυξήσουν τη δυνατότητα ανάπτυξης της δικής τους βιώσιμης ενέργειας, είτε είναι ηλιακή ή η ολική, κυρίως πυρηνική ενέργεια. Και οι χώρες που μέχρι τώρα ήταν πολύ αντίθετες όσον αφορά τη χρήση πυρηνικής ενέργειας, τώρα διρωτώνται, προβληματίσονται. Μήπως πρέπει να γίνουν ανεξάρτητες, ανεξάρτητες από την ε, εφοδιασμό ενέργειας. Και διερωτώ και λέγω, παίζοντας με την ενέργεια για διπλωματικές πιέσεις. Ας αφήσουμε εκτός διαφθορά κλπ. Μήπως αυτό το παιχνίδι έχει συνέπειες σε δεύτερο επίπεδο. Δηλαδή, κάποιοι πολίτες, κάποιοι λαοί, κάποιοι υπεύθυνοι να αρχίσουν να συλλογίζονται. Μήπως μπορούμε να γίνουμε ενεργειακά ανεξάρτητοι με διαφορετικό τρόπο, μέσω τεχνολογίας και έρευνας, για να γίνουμε ανεξάρτητοι. Ίσως η κρίση του φυσικού αερίου αλλάξει την οτροπία. Και μήπως αυτή η αλλαγή νοοτροπίας ε, δημιουργήσει προβλήματα οικονομικά σε εκείνους που προμηθεύουν την ενέργεια. Η πυρηνική ενέργεια καλή είναι, αλλά χρειάζεται και παράδοση ουρανίου, λέει ο Πρόεδρος. Δίκιο έχετε. Αλλάζουν οι παράμετροι. Άλλωστε η θυμή Άλλος τις αγορεύει, βούλετε. Κανείς άλλος. Σχόλια, απαντήσεις από το πάνελ. Θα ακολουθήσουμε αντίστροφη σειρά από τις τις παρουσιάσεις. Ξεκινώντας από τον κύριο Βίλσον. Δεν ετέθησαν άμεσα ερωτήματα αλλά να δώσω σύντομη απάντηση στο ερώτημα του κύριου Τάνοκ περί Ουκρανίας. Βέβαια είμαστε άκρως απογοητευμένοι λόγω της διπλής ηγεσία της Ουκρανίας που η Ουκρανία δεν μπορεί να κινηθεί επί διαφόρων ζητημάτων και η Ουκρανία είναι απογοητευμένη βέβαια αλλά δεν νομίζω θα βελτιωθεί η κατάσταση αντιθέτως. έχουμε θανάσιμη μάχη αν θέλετε κάποιου είδους και η κυρία Τιμοσέγκο κερδίζει λόγω της συμφωνίας που πέτυχε, κερδίζει και στο πολιτικό επίπεδο και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, εξωτερικών σχέσεων. Είναι ο καλύτερος καινούριος και καλύτερος φίλος της Ρωσίας και οικονομικά. Διότι ο αντίπαλός υποστήριξε κύκλους του Προέδρου κλπ. Και αν βγει ο αντίπαλός της εκτός μάχης είναι προς όφελος της. Είναι καλή συμφωνία γιατί Τιμοσέγκο, η Ιουσέγκο θα, θα αντεπιτεθεί γιατί είναι σε, αντίθετη, σε αδύναμη θέση. Το επόμενο εξάμεινο ίσως να δούμε τρελά πράγματα. Όχι μόνο το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας επετέθη κατά του Πρωθυπουργού, αλλά και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή του Προεδρία της κ. Μποροχόφσκα αναφέρθηκε σε ε, προδοσία, έτσι χαλαρά, χωρίς αποδείξεις το Σεπτέμβριο που πέρασε, ο Πρόεδρος ίσως στρέψει την ε, εισαγγελία κατά του Πρωθυπουργού, της Πρωθυπουργού. Και αναφέρονται διάφορα πράγματα, ε, βρώμικα πολιτικά παιχνίδια παίζονται εκεί. Και θα εξακολουθήσουν αυτά μέχρι ότου στις επόμενες εκλογές δοθεί κάποια λύση. Που αν είναι ελεύθερες και δίκες η κυρία Τιμοσέγκο μάλλον θα κερδίσει. thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ, λέει και ο Σποπέσκου. Ετέθησα κάποια πράγματα για την οικονομική κρίση. Να πω κάποια πράγματα λοιπόν και εγώ. Δεν θα ήταν πολύ σοφό να βασίσουμε τη μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη πολιτική μας τώρα βάσει των οικονομικών δυσκολίων που αντιμετωπίζει η Ρωσία σε δύο χρόνια θα ανακάμψει η Ρωσία πιθανότατα και παρά τις κάποιες αλλαγές τόνου και τακτικής της ρωσικής πολιτικής νομίζω ότι η πολιτική που είδαμε τελευταία χρόνια θα παραμείνει και για την επόμενη δεκαετία λίγο πολύ. Η ισχύ της Ρωσία δεν πρέπει να υπερεκτιμάται όπως πριν αλλά δεν πρέπει να υποτιμάται. Επίσης, άρα χρειάζεται στρατηγική εταιρική συνεργασία με τη Ρωσία βάσει εκτίμηση τακτική που ακολουθεί και να λάβουν και όψη για τι συνέπειε οικονομική κρίση. Δεύτερον, όσον αφορά την οικονομική κρίση που έχω να πω. Πράγματι, πιθανότατα θα επηρεάσει και τι γειτονικέ χώρε περισσότερο από ό,τι επηρεάζει την Ρωσία κατά κάτι μέρο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Και αυτό θα έχει και συνέπειε και για την συνεργασία και τελικη σχεση σχέση Ρωσία-Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι είδαμε τα προσφατά χρόνια. Αυτά που συμβαίνουν στη γειτονία, ο πόλεμο στη Γεωργία, η κρίση φυσικού αερίου με την Ουκρανία, είτε και μικρότερε κλίμακα κρίση που συμβαίνουν στη γειτονιά, έχουν και συνέπειε και για την εταιρική σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση Ρωσία. Περιέπλεξαν τη σχέση αυτή. Έχουν εμπλοκαριστεί διάφορα θέματα και υπονομεύτηκαν πυρκύλο τρόπο ε, οι σχέσει αλληλεγγύη με τι ανατολικέ χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανεξάρτητα από τα, αυτά που θα συμβούν με τη Ρωσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, Εξίσου σημαντικό είναι αυτό που θα συμβεί και στη γειτονιά της Ρωσίας. Διότι επηρεάζουν και τους πυλώνες του ευρωπαϊκού προγράμματος αυτά που συμβαίνουν. Οι πολιτικές που ακολουθούν τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν της Ρωσίας και της Ουκρανίας επηρεάζουν την της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επηρεάζουν την ΚΕΠΑ, επηρεάζουν τις προσπάθειες επίτευξης ε, περικοπών σε κομπές διοξιδίου του άνθρακο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την, τον ασφαλή φουδιασμό σε ενέργεια. Και το θέμα περί Ουκρανίας ουσιαστικά δημιουργεί και άλλο ερωτηματικό. Τι είδους γειτονιά θέλουμε να δούμε την επόμενη δεκαετία και πιθανότατα έχουμε τρεις εναλλακτικέ. Πρώτον, ενοποιημένη ζώνη επιρροής της Ρωσίας και σταθεροποιημένη, παγιωμένη και πολύ το υποστήριζουν στη Ρωσία. Δεν είναι το δόγμα Πούτιν με Τβιέντεφ Είναι βαθύτερο το θέμα. Μια δυνατότητα για τη γειτονιά είναι ε, ξαναενοποιημένη ζώνη επιρροής. Δεύτερη δυνατότητα είναι παρόμοια συνεχής κρίσης, ε, προβλήματα που θα επηρεάσουν το πώς βλέπουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ένα το άλλο και πώς θα αναπτυχθεί και τελική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Και η τρίτη πιθανότητα για τη γειτονιά είναι η ανάπτυξη ενός είδους φιλανδικού μοντέλου χωρών που είναι ενταγμένα λίγο πολύ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσεκτική εσωτερική πολιτική, ουδέτερα κράτη-μέλη, βασικά δημοκρατικά και ευρωπαϊκά. Το θέμα είναι ανοιχτό. Πώς θα αναπτυχθεί αυτή η γειτονιά και το πώ θα αναπτυχθεί η γειτονιά θα αποφασίσει ποια θα είναι σχέσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσία και τι μορφή θα έχουν οι σχέσει αυτέ την επόμενη δεκαετία. Ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστώ. Λέω Πρόεδρος, νομίζω ότι η συζήτηση αυτή που έκανε τώρα το δεύτερο πάνελ ήταν και ευρύτερη της Ρωσίας. Πριν ε, δώσω τον λόγο στον... Α, με συγχωρείτε, κάτι ξέχασα, ναι. Α, ξέχασα τον Άντερς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επτά ερωτήσεις τέθηκαν. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Πρώτη ερώτηση Τάνοκ. Εάν ο Ιουσένικο ε, ε, θα προτιμούσε 5 δισεκατομμύρια δολάρια από τη Ρωσία ε, και μίλησε για αυτή την συμφωνία που του θυμίζει το σύμφωνο ριμπεντροπ Ρίμπεντροπ-Μολότοφ. Νομίζω ότι θα το ήθελε. Δεν έχουν οι Ηνωμένε πολιτείε δεν μπορούν να κάνουν τίποτα στην Ουκρανία. Η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μηχανισμού για να συγχρηματοδοτήσει. Πρόκειται για μια χειρονομία που κάνει η Ρωσία απέναντι στην Ουκρανία και είναι επαναστατική και θα πρέπει μάλλον να εκτιμηθεί και όχι να απορριφθεί. δεύτερη ερώτηση του κ. Μπίσλεϊ σχετικά με το ποιες αλλαγές γίνονται τώρα στην Αμερικανική πολιτική. Νομίζω ότι πολλά πράγματα αλλάζουν με τη νέα κυβέρνηση. Αλλάζει η γενική νοοτροπία στην ε, ε, Ουάσιγκτον. Θεωρούν πλέον ότι η ε, πολιτική μπούς απέναντι στη Ρωσία ήταν ανύπαρκτη στην πραγματικότητα. Θα υπάρχει τώρα συντονισμός από το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας, θα ενισχυθεί η θέση του ε, Διευθυντού που ασχολείται με τη Ρωσία στο ε, Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας. Υπό την κυβέρνηση Μπούς η πολιτική, Ρωσία, η πολιτική για τη Ρωσία ήταν κατάλοιπο άλλων πολιτικών, κάτι το οποίο ενοχλούσε τους Ρώσους γιατί θεωρούσαν ότι η αριστερά της Ουάσιγκτον δεν γνώριζε τι ποιος η δεξιά της. Για το ποια θα είναι η νέα πολιτική νομίζω ότι είναι προφανές. Το Ιράν θα είναι πολύ λιγότερο συνδεδεμένο με την ε, Ρωσία και θα είναι καθαρά υπόθεση Ιράν. Με άμεσες ε, επαφές με το Ιράν και το θέμα της ε, αντιπυραυλικής ασπίδας θα διασυνδεθεί με το Ιράν. Το δεύτερο αποτέλεσμα που θα δούμε, πολύ πιθανόν, είναι ότι η νέα κυβέρνηση θα εξετάσει θετικά την Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη Ασφάλειας που ε, προτάθηκε ήδη από το Βερολίνο πέρσι τον Ιούνιο και για το οποίο μίλησε ο Ρώσος εκπρόσωπος Καζετσόφ πριν, γιατί η νέα κυβέρνηση ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο για πολυμερείς συνεργασίες. Ένα τρίτο θέμα είναι ο έλεγχος των εξοπλισμών. Οι συμφωνίες START και ΣΑΛΤ που θα προχωρήσουν τις επόμενες, επόμενα χρόνια πρέπει να αναθεωρήσουν γιατί λήγουν τώρα και η συμφωνία ΚΕΠΑ θα πρέπει να συζητηθεί στην Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη Ασφάλειας. Επίσης η κυβέρνηση Bush δεν είχε δείξει κανένα ενδιαφέρον για τις οικονομικές σχέσεις 38 χώρες στον κόσμο και πολλές από τις ευρωπαϊκές χώρες μέλη έχουν διμερείς σχέσεις για επενδύσεις στη Ρωσία. Η Αμερική δεν έχει. η συμφωνία για την μη στρατιωτική χρήση της πυρηνικής ενέργειας που συνήρθη την προηγούμενη άνοιξη και δεν ε, κυρώθηκε λόγω του πολέμου στην Ρωσία, όλο πρέπει να κυρωθεί και θα έχει σημαντική βαρύτητα. Κανένας δεν είναι αντίθετος, αλλά δεν εντάσσεται τόσο καλά στις ευημερείς Πολλά πράγματα λοιπόν μπορούν να ξεκινήσουν τώρα. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να ερμηνευθεί η δήλωση Biden ότι χρειάζεται μια επανεξέταση των σχέσεων. Δεν σημαίνει όμως ότι θα είναι πιο ήπια η προσέγγιση, η αμερικανική προσέγγιση δηλαδή, αλλά χρειάζεται πιο πολυμερής χαρακτήρας, για παράδειγμα για τα θέματα δημοκρατίας. Και ένα σημαντικό μέρος θα είναι και περισσότεροι συνεργασία με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Η νέα κυβέρνηση Ομπάμα είναι πολύ πιο φιλοευρωπαϊκή. Οι απόψει των ανθρώπων που την απαρτίζουν για την εξωτερική πολιτική δηλαδή είναι τέτοια. Ένα μεγάλο ερωτηματικό είναι αν οι Ηνωμένε Πολιτείε θα θελήσουν να ε, συνεργαστούν για ε, την, ενεργειακή, για την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική. Και ένα άλλο θέμα που θέσατε ήταν ότι μάλλον ο Πούτιν δεν θα αλλάξει τις σχέσεις. Το ζήτημα είναι μήπως οι Ρώσοι αλλάξουν τον Πούτιν. Είναι πιο εύκολο να αντικατασταθεί ο Πρωθυπουργό παρά ο Πρόεδρος βέβαια. Όταν εκλέχθηκε όταν εκλέχθηκε ο, ε, ε, ο πρόεδρος διπλασιάστηκαν κατά κάποιο τρόπο οι ρωσικοί πολιτικοί θεσμοί, γιατί είναι τώρα δύο, και Πούτιν και Μετβιέντεφ. Η Ρωσία είναι βέβαια πάρα πολύ ευαίσθητη σε θέματα διακυμάνσεως των ε, ε, τιμών των πρώτων υλών. Νομίζω ότι κάτι για το μέλλον είναι διαμεσολάβηση. Και γενικά όλο, όλη η πολιτική για την αντιμετώπιση της κρίσης δεν ήταν σωστή. Η ομάδα περί των Πούτιν θεώρησε ότι ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για να μπορέσει να ελέγξει τις τελικές τιμές. Και ο στόχος είναι μην φύγετε τα κακό κείμενα. Μέχρι τώρα η Ρωσία έχει βέβαια τεράστιους πόρους, αλλά δοκιμάζονται τώρα. Και επειδή εξαρτάται τόσο πολύ η Ρωσία από τις τιμές των ποτών θα ανεβοκατεβαίνει η οικονομική της κατάσταση. Ας μην υπερτιμούμε τις αδυναμίες της Ρωσίας, γιατί αυτή η αδυναμία η τωρινή μπορεί να είναι και προσωρινή. Από την άλλη μεριά είναι και μια ευκαιρία για να περάσουμε σε μια κατάσταση όπου η Gazprom θα συμμορφώνεται με τις υποχρώσεις της. Αυτό δεν το ξέρουμε. Έχει έρθει η ώρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητήσει διαφάνεια για την παραγωγή, τα αποθέματα, την μεταφορά του φυσικού αερίου και γνωρίζοντα το τι συμβαίνει γενικότερα και να γνωρίζει γενικά τι συμβαίνει στον τομέα τη ενέργεια στη Ρωσία. Διότι είδαμε την Ευρώπη να, ε, τον Ιανουάριο να, να, να μένει παθητική. Δεν μπορούσα να το φανταστώ. Και πρέπει να επαναξεταστεί η, στάση αυτή. Η Κάσπρομ, βέβαια δεν έχει πόρους ε, για να ε, φτιάξει μόνη της ε, ας πούμε αγωγούς μέχρι την Κίνα θα χρειαστούν πολλά χρόνια αυτό που μπορούμε να ελπίσουμε είναι η Κάσπρομ να επενδύσει αρκετά στο εξορυκτικό πεδίο Αμάλ γιατί όταν πέφτει η ναι. Και νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά είναι αρκετά αμφίβολα σχέδια σε εμπορικό επίπεδο και πρέπει να επιληθούν με άλλες μεθόδους. Εάν η Gazprom δεν επενδύσει λοιπόν για την παραγωγή, όταν αυτά τα τέσσερα πεδία φυσικού αερίου βλέπουν να μειώνεται η παραγωγή τους, ότι θα μειωθεί και η ικανότητα της Gazprom να παραέχει φυσικό αέριο και θα πρέπει να τροποποιηθούν οι προβλέψεις. Το τέταρτο ερώτημα ήταν η επίπτωση της προσχώρησης της Ρωσίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, η γενική εκτίμηση είναι ότι αν η Ρωσία μπει στον ΠΟΕ, θα προσθέσει μισό με 1% στους ρυθμούς ανάπτυξης του εμπορίου, λόγω καλύτερου εμπορίου υπηρεσιών και καλύτερων, μάλλον στο ΑΕΠ της Ρωσίας, λόγω καλύτερων συνθήκων για εξωτερική άμεση επένδυση κατά πόσα πιθανότητα θα αυξηθούν οι τιμές ε, φυσικού αερίου και θα προσεγγίσουν το επίπεδο της παγκόσμιας αγοράς, διότι το επίπεδο της παγκόσμιας αγοράς ούτως ή άλλως έχει χαμηλώσει. Σε ένα-δύο χρόνια λοιπόν θα επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Η ημερομηνία στόχου είναι περίπου το 2011 και αυτό είναι μια θαυμασία ευκαιρία <clears throat> για να υπάρξει εξοικονόμηση ενέργειας για να απαντήσω στο ερώτημα του κυρίου Πρέμπετης και φυσικά όπως λέτε αυτό είναι ένας λόγος να προχωρήσουμε προς διαφοροποίηση της παροχής ενέργειας για να κάνουμε όμως κάτι τέτοιο θα ήταν καλύτερα να υπάρξει πλήρης ενσωματωσία στην αγορά του ενεργειακού τομέα <clears throat> από δεσμοποίηση παραγωγής, από διανομή κτλ. και επομένως να αναγκαστεί και η Gazprom να φιλελευθερωπήσει τις δραστηριότητες. Έχει φιλελευθερωποιήσει μέχρι στιγμής αρκετά και είναι αρκετά διαφοροποιημένη η Gazprom και μέσα στο πλαίσιο αυτό νομίζω αγορές όπως η Σουηδία και η Φιλανδία που έχουν φιλελευθερωποιημένες αγορές είναι πολύ λιγότερο τροτές λόγω αυτού του γεγονότος. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι η φιλελευθερωποίηση της αγοράς ενέργειας θα είναι ο δρόμος με τον οποίο θα προωθήσουμε και μια μεγαλύτερη διαφοροποίηση παροχής, αλλά συγχρόνως θα ήθελα και να τονίσω ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την ενεργειακή χάρτα η οποία δημιουργεί ένα ευρωπαϊκό οργανισμό κοινή δράση για τα ενεργειακά θέματα πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο και σε μια εποχή που η Ρωσία είναι σχετικά ασθενική στον ενεργειακό τομέα, αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή να εμπλέξουμε και να δεσμεύσουμε πλήρως την ε, Ρωσία στην ενεργειακή χάρτα μετά από τις θαυμάσεις εξάλλου δηλώσεις του Πούτιν για την ενέργεια στα πλαίσια της σύγκρουσης για το φυσικό αερίο. Σας ευχαριστούμε κύριε Άσλουντ. Με μεγάλο ενδιαφέρον ακούσαμε αυτά τα οποία είπατε. Ίσως θα μπορέσουμε λοιπόν να αν να υπάρξει να επιτύχουμε την ανάνυψη της ενεργειακής χάρτας, αν η Ρωσία το θέλει και το δέχεται και η Ουκρανία, γιατί όχι, όλα αυτά μέσα σε ερωτηματικά βέβαια. Εν πάση περιπτώσει είναι ο καιρό για να κάνουμε τα τελικά μας σχόλια. Ο κ. Σονισκέβης θα το πράξει αυτό, αλλά προτού του δώσω το λόγο. Σας υπενθυμίζω αυτά που λέει το έγγραφό μας για τη σύσταση προς το Συμβούλιο για τη νέα συμφωνία με τη Ρωσία. Το σχέδιο αυτό ε, σύσταση, είναι μια δεύτερη αναθεωρημένη μορφή. Έχει τροποποιηθεί λόγω των γεγονότων του δεύτερου μισού του 2008 και είχε παγώσει μετά από τον πόλεμο της Ρωσίας-Γεωργίας πριν από τη διαπραγμάτευση, πριν αρχίσει η διαπραγμάτευση τη νέα συμφωνία, οπότε με την απόφαση να αρχίσουν και πάλι διαπραγματεύσεις το 2009, βγάλαμε από την κατάψυξη το έγγραφο αυτό. Ο κύριος Ονισκέβιτς κάνει με ορισμένε προτάσεις σε σχέση με αυτό το έγγραφο και ζητάει να υπάρξουν βελτιώσεις ποιοτικού χαρακτήρα σε σχέση με την τωρινή συμφωνία εταιρικού και εμπορικού χαρακτήρα και ζητά να ενισχυθούν στοιχεία όπως δημοκρατία, το σεβασμό του κράτους δικαίου, σεβασμός για θεμελιώδεις ελευθερίες και ανθρώπινα δικαιώματα και άλλα πολλά. Προθεσμία για τροπολογίες. 20 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι όλες οι τροπολογίες που έχουν κατεθεί στο προηγούμενο κείμενο 11 Σεπτεμβρίου του 2008 έχουν εκπέσει. Η νέα καταληκτική προθεσμία είναι 20 Φεβρουαρίου το μεσημέρι. Ε, να και λοιπόν στα μέλη της Επιτροπής μας να σκεφτούν αν θέλουν να καταθέσουν τροπολογίες ή όχι. Έχουμε ακόμα μία εβδομάδα μπροστά μας. Κύριε Ονισκιεβίτς, σας παρακαλώ, παρακαλώ να συνοψίσετε αυτή την τόσο πλούσια συζήτηση τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο πάνελ. Ευχαριστώ. Δεν είχε τη μορφή διαπραγματεύσεων η συζήτησή μας, άρα δεν θα μπορούσα να πω πολλά επί των όσων συμφωνήσαμε, αλλά κάποια γενικά σχόλια νομίζω ότι θα ήταν ενδεδειγμένα. Το πρώτο σχόλιο μου είναι ότι η φύση των σχέσεών μας με τη Ρωσία, πια είναι, όλοι συμφώνησαν ότι αυτοί, αυτές οι σχέσεις είναι ζωτική σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση το θέμα είναι θα πρέπει να τις αποκαλέσουμε στατηγικές σχέσεις ή εταιρικέ. Αυτό είναι θέμα συζητήσιμο. Στατηγικές σκέψεις, σχέσεις συγγνώμη, θα έδειχναν πόσο σημαντικές είναι οι σχέσεις, πόσο σημαντικό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει ε, πάνω σε κάποια σημαντικά στατηγικά ζητήματα, αλλά η εταιρική σχέση συνεπάγεται κάποιε κοινέ αξίε και αυτό είναι κάτι που αμφισβητείται κατά πολύ από εμά κατά πόσο έχουμε κοινέ αξίε. Κυρίω λόγω τη φύσεως του ρωσικού πολιτικού συστήματο που πολλοί θεωρούμε ότι δεν είναι μια πλήρω ελεύθερη δημοκρατία αλλά ένα νέο είδους δημοκρατία χαλιναγωγούμενη δημοκρατία κυρίαρχη δημοκρατία δεν ξέρω έτσι αποκαλείται sovereign democracy στη Ρωσία κυρίαρχη δημοκρατία ε, παραμένει εξαιρετικά σημαντική η Ρωσία για μας, για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι η ενέργεια. Δεν θα ήθελα όμως να συνοψίσω τα ήδη λεχθέντα. Θα ήθελα να αφαιρθώ σε κάποια άλλα ζητήματα που εθίγησαν. Πρώτα απ' όλα εκτίμησα πολύ τη δήλωση του κύριου Κοσατσόφ ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει όλα τα ευρωπαϊκά κράτη ισότιμα, αλλά στην πράξη βλέπουμε τα πράγματα ότι είναι διαφορετικά. Δυστυχώς να επενθυμίσω αυτό που πολύ συχνά έλεγαν Ρώσοι πολιτικοί για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έλεγαν ότι το είναι καλύτερα να συνομιλεί κανείς διμερός διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασικά είναι ανε, αργή. Άρα μερικά πράγματα καλύτερα ρυθμίζονται διμερός και ελπίζουμε ότι αυτές οι μεγάλες χώρες θα προωθήσουν τα πράγματα πιο γρήγορα και λιγότερο πειθαρχημένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα ακολουθήσουν. Μάλλον λιγότερο πειθαρχημένες θα έχουν την τάση να έχουν αντίρρηση. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και ερχόμαστε στο πρόβλημα της αλληλεγγύης που το έθεσε σαφώς ο κ. Βίλσον και ο κ. Πάσκο που είναι σημαντικό για την συνοχή και αποτελεσματικότητα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε επίσης και το θέμα που είναι πολύ βασικό. Είχαμε φιλόδοξο πρόγραμμα να δημιουργήσουμε τέσσερις κοινούς χώρους με τη Ρωσία. Ένας από τους χώρους που υποτίθεται θα οικοδομούσαμε με τη Ρωσία ήταν κοινό χώρος ασφαλείας. Κυρίως λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις στη στην ε, Γεωργία και στην Απχασία. Δεν ξέρουμε αν αυτό είναι κάτι βιώσιμο που προγραμματίζαμε ή αν θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σύστημα τύπου ΟΑΣΕ ή να δημιουργήσουμε στην Ιρλανδική Χάρτα για τη Νέα Ευρώπη και διάφορα συναφή. Και για να μην μακρηγορήσω, όσον αφορά τα συμπεράσματά μου, να παραθέσω αυτό που είχε γραφεί στην αρχή των εστώτος έτους από τον Σερ Ρόντρικ Κλάιν, τον πρώην Βρετανό πρέσβη στη Ρωσία, σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε σε ένα έντυπο το οποίο εκδότης είναι ο Σκιούς Λουκιανόφ, το Russian Global Affairs, το συστήνω ένθερμα σε όλους και το άρθρο έχει τον τίτλο «Η Ρωσία και η Δύση είναι αναπόφευκτη αντιπαράθεση» και θα ήθελα να κλείσω παραθέτοντας από το άρθρο αυτό που το, με το οποίο συμφωνώ και έχει ως εξής η παράθεση και παραθέτω προσπαθούμε να είμαστε εταίροι και σύμμαχοι αυτό τελικά δεν ήταν ρεαλιστικό, αποτύχαμε για την ώρα, όμως αυτό δεν θα πρέπει να μας καταστήσει εχθρούς. Πολλά διακυβεύονται και έχουμε πολλά κοινά. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ κύριε Νισκίεβιτς. Δεν ξέρω πόρα αυτό που είπατε αν ήταν πιο πολύ πικρό ή πιο πολύ ε, αισιόδοξο μήνυμα. Πάντως η πιο πολυ αισιοδοξο ήταν εξαιρετική και από την σκοπιά των μελών και ευχαριστώ ιδιαίτερα όλους τους παρεμβάντες, τον κύριο Κοζατσόφ, πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Θεμάτων της ε, Δούμα, τον κύριο Λουκιάνοφ, αρχισυντάκτη αυτού του εξαιρετικού περιοδικού, τον κύριο Μόσες ε, του Φιλανδικού ε, Ιδρύματος Ινστιτούτου για Εξωτερικές Σχέσεις, τον κύριο Άσλουντ, τον εμπειρογνώμονα από το Πέτερσον, τον κύριο Λούνσεν και Ποπέσκου, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων. Ευχαριστώ και διακόπτη συνεδρίαση.